Colleagues, if you could take your seats. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Yeah. Okay. First of all. Ωραία λοιπόν. Καταρχάς, συνάδελφοι, να εγκρίνουμε το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της συνεδρίασης της 5ης και 6ης Νοεμβρίου. Υπάρχουν ενστάσεις, αν όχι, εγκρίνονται. Να περάσουμε λοιπόν στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων με το συντονιστή για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Έχουμε τέσσερις συντονιστές σήμερα και 5 αύριο το απόγευμα και χαίρομαι που έχουμε ξανά εδώ την Κάρλα Πέις διότι είναι πάντα ευχάριστο να καλωσορίζουμε πρώην συναδέλφους. Ξέρω ότι έχετε ε, αρμοδιότητα για τα προγράμματα προτεραιότητας 18 και 30 το πρόγραμμα 30 για το Σικουάνα Σέλτ. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας δίνω το λόγο για 10-15 λεπτά και από εκεί και πέρα θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Ε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε 10 λεπτά για κάθε συντονιστή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η χρονιά αυτή ήταν μεταβατική για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων. Εδώ και πολλά χρόνια είχαμε διάφορες μελέτες, τις οποίες υποστήριζε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγιναν μελέτες σκοπιμότητας, Η αξιολόγηση έγινε και για του πιο σημαντικούς αυτούς δύο διαδρόμους και τα σημεία που έχουμε συμφορήσει και τα προγράμματα προτεραιότητας 18 ε, και 30 γίνονται για να έχουμε σύνδεση ε, στις βασικές λεκάνες από το Σικουάνα και το Μεΐσι ε, και από εκεί και πέρα από την Πενελούξ στη νοτιοανατολική Ευρώπη και να φτάσουμε μέχρι και μέσω των ποταμών επικοινωνίας μέχρι τον Εύξηνο Πόντο. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η νότια συνεργασία με περιβαλλοντικές ομάδες. That was helped by the... Και είχαμε και την ολοκλήρωση της κοινή δήλωση των κατευθυντηρίων γραμμών για την εσωτερική ναυσιπλοεία και ε, τη ε, διευρωπαϊκά δίκτυα μας ενδιαφέρει και η ανάπτυξη της ναυσιπλοεμίας αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος και των οικοτόπων που έχουμε ε, εκεί και θέλουμε να επιτύχουμε και τα δύο. Πάντα μας απασχολούν και τα δύο και μα ενδιαφέρει και η αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θέλουμε να μελετήσουμε και αυτά. Υπάρχει και μια αξιολόγηση, από εκεί και πέρα είδαμε και τη στρατηγική για το Δούναβι. Αυτή η στρατηγική ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010, φαντάζομαι ότι θα το γνωρίζετε όλοι αυτό. Και από εκεί και πέρα είχαμε και ε, μια έκθεση για την ανάπτυξη των διαδρόμων προτεραιότητας, ε, και μας ενδιαφέρουν και τα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας εδώ. Έχουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα της ανάπτυξης ε, ε, του Σικουάνα στη βόρεια πλευρά και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν διάφορες ε, διαδικασίες. Έχουμε συμφωνία τώρα μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας και επισημάνεται το γεγονός ότι οι ποταμοί δεν αποτελούν μόνο ευκαιρία για τις ε, ε, μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοείας, αλλά είναι καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη των, ε, των γειτονικών περιοχών και την επίλυση και άλλων σχετικών προβλημάτων. Βέβαια τα πάντα δεν ήταν ομαλά στη διάρκεια του προηγούμενου έτους λόγω των οικονομικών δυσκολιών που έπληξαν τις περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχουν ε, προβλήματα με την ε, επενδύσεις και την νέα ανακατανομή των πόρων και αυτό φυσικά είχε και αρνητικές επιπτώσεις σε ισχυρό βαθμό στην περιοχή του Δούναβη. Για το πρόγραμμα προτεραιότητας 18 τώρα, που είναι η σύνδεση μεταξύ των εσωτερικών περιοχών στο Δούναβι. Εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ο κύριο Κάλλα, ο Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπήρχε ένας Ευρωπαίος συντονιστή και διοργανώθηκε μια συνάντηση των ε, Υπουργών Μεταφορών ε, στο Λουξεμβούργο το Δεκέμβριο του 2011 και εκεί συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχουμε και πώς μπορούμε να τα λύσουμε αυτά στο μέλλον. Και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και κάποια αξιοπιστία προς τις επιχειρήσεις για τα θέματα των μεταφορών, γιατί αυτό μας απασχολούσε τότε. Ε, εκείνο το οποίο κατέστη σαφέ είναι ότι χρειάζεται πολιτική δέσμευση για να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα τα οποία μα αφορούν στο Δούναβι, καθώ επίση και ε, την πτυχή τη ανάπτυξη, ε, τι επιπτώσει για το περιβάλλον, ε, κατάλληλη διαχείριση των υδάτων, καθώ επίση και ανάπτυξη ε, κέντρων επιμελητίας, κυρίως ε, λιμένων και ε, προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν τις τοπικές οικονομίες των χωρών που τις αφορά το πρόγραμμα αυτό. Τώρα, για τα διασυνοριακά τμήματα και τα βασικά προσκόμματα που υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση. Το πρώτο βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε είναι το τμήμα του Δούναβη μεταξύ Στρασβούργου και της ε, Βαβαρίας. Η μελέτη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το τελικό σχέδιο έκθεσης βρίσκεται ε, στα χέρια του Ομοσπονδιακού Υπουργείου και θα παρουσιαστεί στις 22, παρουσιάστηκε συγγνώμη, στις 22 Νοεμβρίου και από εκεί και πέρα θα χρειαστούν μερικοί μήνες ακόμα μέχρι η ομάδα παρακολούθησης να ολοκληρώσει τις εργασίες της. Από το σχέδιο κειμένου που είχαμε και την τελική ανάλυση αναφέρεται ότι υπάρχει πρόβλημα και στις δύο περιπτώσεις. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στις υποδομές και έχουμε μια ανάλυση κόστος εφολίας που φτάνει στο 6,5%. Μας ενδιαφέρουν επίσης και οι υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες για να έχουμε ε, αξιόπιστες ε, συνθήκες ναυσιπλοέας και θα πρέπει να ανάλυση κόστος ωφελίας στις τάξεις του 7,6%. Όλες αυτές οι πληροφορίες βέβαια θα δοθούν ε, στις αρχές του νέου έτους και θα συζητηθούν περαιτέρω. Και αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει και μια σχετική διάσκεψη που θα συζητήσει το θέμα αυτό. Μετά, έχουμε την Ανατολική περιοχή της Βιέννης. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα επιτυχημένης ιστορίας το πρόγραμμα είχε σταματήσει για πάνω από δύο χρόνια για τις παρεμβολαντικές έρευνες, αλλά την περασμένη εβδομάδα έγινε μια ανάλυση από τη ΒΒΕΦ και η ΒΒΕΦ είπε ότι το πρόγραμμα αποτελεί βέλτιστη πρακτική και αυτό ε, θα έχει θετικές συνέπειες αν εφαρμοστεί και σε άλλους ε, ποταμούς. Ε, διατηρούνται υψηλά επίπεδα και γίνεται αξιολόγηση βαθμιδών όπως προχωράει η διαδικασία. Ε, στο βουλγαρικό τώρα τμήμα, η μελέτη για τη βελτίωση της ε, ναυσιπλοείας στο βουλγαρικό τμήμα ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2011, ακριβώς δηλαδή πριν από ένα χρόνο και από εκεί και πέρα οι άδειε για να προχωρήσουμε στο δεύτερο τμήμα των ε, κατασκευών σταμάτησαν από τις αρχές της Ουγγρικής κυβέρνησης γιατί ε, θεωρήθηκε ότι δεν συμμορφούνται με την κείμενη νομοθεσία. Και ε, το δικαστήριο του Δήμου του Κάσκη θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να αναπτυχθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ουγγρική κυβέρνηση να ζητήσει από τους εμπειρογνώμονες να εξετάσουν το πρόγραμμα και να προσπαθήσουν να επιλύσουν αυτή τη διαφορά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα βεβαίω, διότι έκτοτε στη Βουλγαρία υπάρχει τεράστια τεκμηρίωση και στην Ουγγαρία δεν είναι πολύ εύκολο να εξετάσουν ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Εγώ επισκέφτηκα επίσης και τον ε, κοινό τομέα Κροατία-Σερβία και έγιναν κάποιες συζητήσει για να υπάρξουν διμερεί συμφωνίε και εκεί. Για την ε, περίπτωση τώρα Βουλγαρίας-Ρουμανίας υπάρχει ένα μνημένο συνενέωσης για την ανάπτυξη ε, κοινού προγράμματος και υπεγράφει αυτό στη Σόφια τον Οκτώβριο μαζί με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των μεταφορών Και αυτό θεωρώ κατά την άποψή μου ότι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της εσωτερικής ναυτιπλοεία, διότι δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των υδάτων, ε, μπορούμε να δούμε και την, ε, τα θέματα γεω, τα τα θέματα της άρδευση και ούτω καθεξής, ε, τη σεβασμό του περιβάλλοντος, να μειώσουμε το, την αύξηση των οδικών μεταφορών και να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση και να υπάρχουν και καλύτερες ε, ε, πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των ε, περιοχών που βρίσκονται τοπικά. Τώρα, στην περιοχή Βουλγαρίας-Ρουμανίας έχει ξεκινήσει μια σημαντική διαδικασία και μετά από τις υποδείξεις που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο Αναυσιπλοείας ξεκίνησαν κάποια προγράμματα και θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες εξετάζεται και τι γίνεται με τη μετανάστευση και την ε, περίοδο αναπαραγωγή των ε, ψαριών των ποταμών και αυτά θα παρακολουθούνται στενά ε, και θα βλέπουμε τι γίνεται στους τόπους. Έγινε ένα πρώτο εργαστήριο πέρσι με πολύ μεγάλη συμμετοχή ενδιαφερομένων. Αυτά λοιπόν για το πρόγραμμα 18 και τώρα να δούμε το πρόγραμμα 30. Το πρόγραμμα 30 ενώνει την ε, λεκάνη του Σικουάνα βόρεια του Παρισιού με τον ε, ε, ποταμό Σέλτ του Βελγίου. Έχουμε σημαντική σύνδεση και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της περιοχής ενώνουμε τη Βόρεια Γαλλία ε, με μεγάλα θαλάσσιους λιμένες. Ε, έχει προχωρήσει ο διάλογος, αλλά η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα γίνει αναθεώρηση από οικονομική σκοπιά του προγράμματος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τα οικονομικά προβλήματα αυτής της περίοδου. Και φυσικά όλοι επεσήμεναν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό και ε, οι κάτω χώρες υποστηρίζουν την ολοκλήρωση των εργασιών. Ωστόσο όλοι κατανοούν ότι η νέα γαλλική κυβέρνηση ε, πρέπει να κάνει μια νέα ανάλυση και επανεξετάζει τα της χρηματοδότησης, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης στη Γαλλία. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες, οι οποίες όμως δεν υπήρχαν στο παρελθόν Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε και υψηλέ προσδοκίε για να έχουμε θετικά αποτελέσματα εν τέλει και ελπίζω ότι θα βρεθεί μια καλή λύση ε, κατά πάσα πιθανότητα μέσω του νέου μέσου των ομολόγων έργου. Τώρα, στη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Ανατολικής Φλάνδρας και κάτω χωρών για την ανάπτυξη ε, διαδρόμου και εκεί θα είναι πολύ σημαντικό και με την ανάπτυξη του, ε, ε του διαδρόμου Σικουάνα Σέλτ. Υπάρχουν και δραστηριότητες σε άλλες χώρες ε, για την εσωτερική ναυσοσυπλοεία. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Ιταλία υπάρχει ένα πρόγραμμα ε, για το Μπάδο στη Μάντοβα. Ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό χωρίς καμία στήριξη και από εκεί και πέρα υπάρχει ε, στήριξη κατά 10% από την Αρμόδια Επιτροπή προχωράει το πρόγραμμα και εξετάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και για το πρόγραμμα αυτό. Ε, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το πρόγραμμα αυτό, διότι είναι ιδιαίτερη ε, μεγάλη συμφόρηση στην περιοχή αυτή. Θα ήθελα να τονίσω τώρα τα εξής. Αυτό το οποίο επιθυμούμε για το μέλλον είναι καλύτερη ολοκλήρωση των ε, ε, μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοείας με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς ε, και α, καλή οργάνωση των διαδρόμων και χρήση πολλαπλών μέσων μεταφοράς. Δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι μεταφορές στην εσωτερική ναυσιπλοεία, θέλουμε και ανάπτυξη εδαφική των περιοχών και να υπάρχουν και δυνατότητες ε, ανάπτυξης στρατηγικής του Δούναβη. Πραγματικά λοιπόν θέλουμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να επιλύσουμε τα προβλήματα στις περιοχές αυτές. Επιθυμούμε εδρωμένη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων και των περιβαλλοντικών ομάδων και όσο καλύτερη είναι η συνεργασία πριν ξεκινήσουν οι εργασίε, τόσο πιο ομαλά θα προχωρήσουν οι εργασίες ε, στη συνέχεια, αν τουλάχιστον υπάρχει συνεννόηση ω προς τα έργα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν και θα είναι τα πάντα πιο εύκολα για όλους, ε, ώστε να μην υπάρχουν εντάσεις ε, κατέρωθεν. Τώρα, είναι πολύ σημαντικά τα ομόλογα έργο, ιδίω τώρα που βιώνουμε χαλεπούς καιρούς, για τη χρηματοδότηση των ε, προγραμμάτων και κατόπιν υπάρχει και το θέμα των τεχνολογικών εξελίξεων που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Υπάρχουν οι στόχοι του ορίζοντα 2020 Και βεβαίω δεν επαρκούν αυτά. Χρειαζόμαστε νέου κινητήρε, ε, καλύτερα καύσιμα, ε, όπως για παράδειγμα υγροποιημένο φυσικό αέριο και ε, ομαλή λειτουργία όλων αυτών. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε είναι να υπάρχει υποτιλητική στήριξη, καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση των σκαφών, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε σε όλους όσους ζουν ε, στις όχθες των ποταμών ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι τα ε, σκάφη που χρησιμοποιούνται για τις ποτάμιες μεταφορές δεν συνεισφέρουν στην περαιτέρω ρήπανση. θα πρέπει από εκεί και πέρα να υπάρχει μεταφορά στις ε, κατάλληλες αγορές και να υπάρχει και πολιτική βούληση να βοηθήσουμε τους τοπικούς πληθυσμούς. Αν δεν μπορέσουμε να τους αποδείξουμε ότι έχουμε ωφέλη και για αυτούς, τότε δεν θα επιτύχουν τα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή έξι έχουν ζητήσει να παρέμβουν. If we... Αυτή και αν καταφέρουμε Mr. ο κύριος Γκρός επίσης αν ο καθένας περιοριστεί σε δύο λεπτά θα μπορούμε να έχουμε απαντήσεις στις παρεμβάσεις σας και να τηρήσουμε και το στενό περιοριστικό αυστηρό χρονοδιάγραμμά μας. Ο κύριος Ρίκε, δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Ήθελα να ρωτήσω την, τη συντονίστρια για τις διάφορες πτυχές του περιβάλλοντος στον άξονα του Δούναβη και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συντονιστούν αυτές οι πτυχές δεδομένων των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί και επισημανθεί πλημμύρες και το καθεξής. Και δεύτερον, θεωρεί η συντονίστρια ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα με το έργο 30 του ΜΕΦΣΙ, 30 συγκεκριμένα, που είναι σημαντικό πιστεύω προς τον ε, άξονα Δύσης Ανατολής και εάν έχει ασχοληθεί με τα ομόλογα έργου. Η συντονίστρια που είναι πολύ σημαντικό μέσο και ιδιαίτερα σημαντικό για το μέσον. Επίσης δεδομένων των ε, προθεσμιών για τη θεωρητική υλοποίηση των μέσων αυτών η αναθεώρηση των δαπανών είναι πιστεύω πολύ σημαντική. Πρέπει να γίνει. Γιατί έχουν περάσει τουλάχιστον 10 χρόνια που ορίστηκαν αυτέ οι δαπάνε. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν για τα έργα 18 και 30 να γίνει τουλάχιστον γι' αυτό αναθεώρηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρικέ, ήσασταν και σύντομο. Ο κύριο Αλκαντράου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τη συντονίστρια για την, για την ε, παρουσίαση αυτή. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι έχουν ε, παρισφρήσει αρκετές καθυστερήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης τα έργα. Έχουμε λοιπόν μεγάλους άξονες. Και δεν θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τον προγραμματισμό των μεγάλων ε, αξώνων, ιδιαίτερα για το Σικουάνα Έσχη, που προβλέπετε ότι θα καθυστερήσει λίγο περισσότερο από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί. Από πλευρά της Γαλλίας ήδη σημειώνονται καθυστερήσεις. Έχετε λοιπόν κάποιες ε, πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Για τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί στα σύνορα Γαλλίας-Βελγίου. Έχετε πληροφορίες? Δεύτερη ερώτηση. Για να συνεχίσω στο είπε και ο κύριος Ρικέ για τα ομόλογα έργου. Γνωρίζουμε ότι έως το 2014 τουλάχιστον θα είναι περιορισμένα τα κονδύλια. Καλό λοιπόν θα ήταν να προβλέψουμε, να δούμε λίγο τις εξελίξεις πολλά συζητιούνται. Ε, στην πράξη όμως υπάρχουν εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει λοιπόν κάποιο ρεαλιστικό σενάριο που να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση αυτών των μεγάλων έργων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα είμαι και εγώ σύντομη. Γενικά στα διευρωπαϊκά δίκτυα το είπατε κυρία Ταΐσε, οι πλωτές οδοί έχουν συμπεριληφθεί και αυτό επιτέλους τώρα έπρεπε να γίνει αυτό διότι είναι πολύ σημαντικό για περιβαλλοντικές μεταφορές. Έχω τι εξή ερωτήσει. Είπατε ότι στο Στράουμπινγκ ε, για τη μελέτη, για τη στενοπό, δεν είναι αδιαμφισβήτητο. Ποιε δυνατότητε βλέπετε εσεί ε, με την οικονομική κατάσταση να αρθεί αυτή η στενοπό. Δεύτερον, στρατηγική για τη λεκάνη του Δούναβη γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι γενικά η πλοημότητα του Δούναβη, εκεί όπου είναι σκόπιμο και εφικτό περιβαλλοντικά, θα πρέπει να, και να μπορέσει να προαχθεί. Το βλέπετε κι εσείς έτσι. Ποια δυνατότητα υπάρχει να προαχθεί έτσι αυτό. Τρίτη δυνατότητα, ομόλογα έργου. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζω είναι συγκεκριμένα για τις ε, πλωτές οδούς, ε, ποτάμιες οδούς. Υπάρχει κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα που θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2013, δηλαδή για να δούμε κατά πόσον οι πλωτές μεταφορές, ε, ποτάμιες μεταφορές μπορούν να συνενταθούν. Τηρήσατε το χρόνο σας ο κύριο Κράμερ τώρα δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Αλλά μου λείπει κάπως η αξιολόγηση της εσωτερικής ποτάμιας ε, μειώθηκε 20% τα τελευταία χρόνια. Οι εξελίξεις που είχαν προβλεφθεί δεν έγιναν έχουμε στο, στη διόρυγα Ρήνου Δούναβη μόνο 20% των εσόδων. Δεν υπάρχουν πλέον πλοία που να κινούνται στο Δούναβη. Τα προβλήματα που αναφέρετε θυμάμαι πριν από 30 χρόνια ο Κόνραντ Λόρεντς είχε διαμαρτυρηθεί γιατί είχε πει ότι ήταν ανεύθυνο αυτό και το σταμάτησε η αυστριακή κυβέρνηση. Πώς μπορείτε να είσαστε λοιπόν αισιόδοξοι ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και για το Στράουμπινγκ, ο ίδιος ο υπουργό Περιβάλλοντος της ΤΣΕΣΟΥ, χριστιανοκοινωνιστής της Βαβαρίας, είπε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα. Τώρα, αυτό θα μπορούσε να ήταν λογικό στο Ρήνο με μια φιλοπεριβαλλοντική δυνατότητα μεταφοράς. Όχι όμως για, την, για επέκταση για ένα ή δύο πλοία μόνο. Αυτό βλέπω να λείπει στη δική σας αξιολόγηση. Δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς και να έχουμε ευχολόγια. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Για το, ε, τη διόρυγα Rhein-Main-Δούναβη ήταν μια καταστροφή χρηματοοικονομικά για τη Γερμανία. Τελευταίο σημείο, ομόλογα έργων. Δεν υπάρχουν χρήματα. Διαρωτώ με, ποια προγράμματα μπορείτε να προτείνετε όπου θα μπορούσαμε να, εδρασ... να μπορέσουμε να στοχεύσουμε σε αυτά η, ο Σκάλδης μπορεί να ήταν ε, σκόπιμο αυτό. Όλα αυτά δεν θα έθεταν προβλήματα, αλλά για το Δούναβι με 30, 30 χρόνια που συζητάμε για αυτό το θέμα και δεν γίνεται τίποτα. Τελευταίο σημείο, θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι κάπου θα μπορούσε να υπάρξει μια εξαίρεση για την κατηγορία 4 με ε, βάθος τρόπιδας 2,5 ε, εκτόπισμα 2,5 μέτρα βήθισμα. Πώς θα μπορούσατε να το φανταστείτε αυτό. Ευχαριστώ. Να τηρείτε το χρόνο παρακαλώ. Φαντάμ δύο λεπτά κι εσείς. Πρόεδρε ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα θερμά την κυρία Πέις για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει. Δύο λόγια θέλω να πω και για τη χρηματοδότηση και μια παρατήρηση ή παρατήρηση από πλευράς μου επενδύσεις στις υποδομές ε, των ποτάμιων πλώιμων μεταφορών είναι κάτι το ευνοϊκό, αλλά πρέπει μακροπρόθεσμα να υπάρξει δυνατότητα απόσβεσης όλων αυτών των επενδύσεων. Και οι πολιτικοί τίνουν ε, κοντόθωρα σε βραχυπρόθεσμα να σκέφτονται. Αν όμως το δει κανείς σε ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο, τότε θα μπορούσε να είναι κερδοφόρο να κάνουμε επενδύσεις ε, στην ποτάμενα ψηπλοεία για την δική μας ε, περίπτωση της χώρας μας, για τη διόρυγα του ε, βασιλέα ε, Γουλιέλμου του Πρώτου. Βλέπουμε ότι πολλά γίνονται σε, αυτό, σε αυτή τη διόρυγα και πολλά εισπράττει το Ολλανδικό κράτος μέσω των επενδύσεων που έγιναν τότε, μέσω των δράσεων ενός συνετού βασιλιά που μπόρεσε να κοιτάξει προς το μέλλον και να ε, δει τα πράγματα σωστά. Η αναλογία κόστους-οφέλους ε, πρέπει να είναι σωστή. Είπατε κυρία Πάης ότι υπάρχουν τα θέματα των, ε, της χρηματοδότησης. Υπάρχει η ευνοϊκή αυτή χρηματοδότηση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ ήθελα να πω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και να αναφερθώ στο πρόγραμμα, στο σχέδιο του Δούναβη. Επί, ε, πολύ σοβαρά υπήρξε η επίπτωση ε, για την αυσιπλοεία στο Δούναβι με τα προβλήματα που υπήρχαν. Καλωσορίζω την ε, πρωτοβουλία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας πρόσφατα πριν από κάποιες εβδομάδες για τη βελτίωση της ναυσιπλοείας στο Δούναβι και πιστεύω ότι οι πλωτές μεταφορές στο Δούναβι μπορούν να υλοποιούνται και να προχωρήσουν σεβόμενοι πάντα τις αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας. Και σε εκείνες τις ατυχείς περιπτώσεις όπου ε, πλήγει η φύση λόγω τέτοιων ε, προγραμμάτων σε σχέση με τις υποδομές, αυτό δεν πρέπει να παρακολεί άλλα κράτη να αναπτύσσουν εκείνα αυτού του είδους τις μεταφορές σεβόμενα τις υποδομές. Γι' αυτό είμαι ε, ένθερμα υποστηρίζω ε, την προαγωγή των μεταφορών στο Δούναβι με τρόπο που πιστεύω ότι θα σέβεται το περιβάλλον. Για τη διασύνδεση του Ρήνου και του Δούναβη θα έπρεπε να συνεχιστεί το πρόγραμμα ΝΑΙΑΣ ε, στην περίοδο 2014-2020. Θέλω να σας ρωτήσω, θα προαχθεί μια ευρωπαϊκού επίπεδου στρατηγική, ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε από κοινού την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτυχθεί αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική όσον αφορά τις ε, εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ποτάμιες μεταφορές. Εσείς παρακαλώ δύο λεπτά. Καλή σας μέρα κυρία Πέις. Ευχαριστώ για την έκθεσή σας, την εισήγησή σας. Κυρία Πέις, πέρυσι σχεδόν την ίδια ερώτηση είχα διατυπώσει. Πρόκειται για το εξής, για το κομμάτι που αφορά τη Βαβαρία από το Straubing Και πραγματικά ετέθηκε το ίδιο ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν δόθηκε απάντηση ή ανεπαρκή απάντηση δόθηκε. Συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτή η εναλλακτική διαδρομή, αυτή η εναλλακτική δυνατότητα. Μια συγκεκριμένη ερώτηση. Θα το επιτρέψετε οι περιβαλλοντικέ ενώσεις ε, να μπορέσουν ε, να έχουν ένα ανεξάρτητο επαΐοντα που θα αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις επιτόπου. Ναι ή όχι. Και πάντα σε σχέση με αυτά τα θέματα προγράμματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής πότε, ποια προγράμματα θα ξεκινήσουν ε, ίσως θα μπορούσε να υπάρξει ένας χάρτης όπου με διαφορετικά χρώματα να δείχνεται πόσα πλοία κινούνται καθημερινά σε ποιο κομμάτι για να ξέρουμε μεταξύ Στράουμπινγκ και του επίμαχου αυτού τμήματος ε, υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία πλέον από άλλα τμήματα. Παραμένει η ερώτησή μου και θα ήθελα να είχα απάντηση σε αυτήν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος Αλεξής σημαντικός ο κύριος Γκρός. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφε Τάισεν, ευχαριστώ για την εισήγηση. Δεν τα παρακολούθησα, δεν τα άκουσα όλα, αλλά πολλά. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Πολλέ φορές ε, συζητούμε την ανάλυση κόστους ωφέλους. Αυτό είναι ένα κριτήριο που αφορά πολλά προγράμματα που εδώ και πάνω από 10 χρόνια έχουμε εδώ και εξετάζουμε και από τότε που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και διαρκώς ε, βρισκόμαστε στο πεδίο έντασης μεταξύ αποτελεσματικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος και από την άλλη πλευρά δημιουργίας ενός πλήρους δικτύου μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ερώτηση. Σε σημαντικούς τέτοιους άξονες μπορούν να υπάρχουν τέτοιες αναλύσεις κόστου, κόστους-οφέλους. Να ξέρουμε ποια θα είναι τα κόστη, Ποια θα είναι τα ωφέλη μακροπρόθεσμα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Δεύτερον, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις ε, που θα πρέπει να τηρηθούν περιβαλλοντικά. Θα υπάρξουν στενοποί, στενοποί που ε, ανάντι ή κατάντι σε σχέση με κάποια τμήματα θα επηρεάσουν αυτά. Σε σχέση με τις επενδύσεις είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό. Δεν έχει νόημα να πούμε θα επενδύσουμε σε ένα τμήμα τόσα εκατομμύρια όταν ξαφνικά υπάρχει και ένα, μια στενοπός που δημιουργείται σε αυτό το τμήμα. Μια ερώτηση και αυτή αφορά την επόμενή σας ίσως επίσκεψη. Δεν θα είναι η τελευταία σας επίσκεψη. Ποια είναι η πρόταση που συνδέει τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με τις ε, μελλοντικές. Υπάρχει συνοχή και συνεκτικότητα. Εγώ πιστεύω ναι, αλλά θα υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις ή διορθώσεις που θα έπρεπε να γίνουν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Προτού απαντήσετε Κάρλα σε αυτά, είναι κρίμα το ότι δεν μπορούμε να δούμε πώς ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαμε να έχουμε νερό που θα περάσει μια και εκεί δεν έχουμε σίγουρα ξηρασία με τις πλημμύρες και όλα που έχουμε για να ανακουφιστεί η περίπτωση αυτή και σε σχέση με το Δούναβι. Έχετε τον λόγο Κάρλα για να απαντήσετε παρακαλώ. Ναι, θυμάμαι μια συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο όπου είχε προταθεί να μεταφερθούν να μεταφερθεί νερό από την Αυστρία στην Ισπανία, το θυμάστε, με ένα μεγάλο αγωγό. Αλλά τελικά οι Αυστριακοί δεν ενθουσιάστηκαν πολύ. Δεν ήθελαν να στείλουν το νερό του στην Ισπανία. Αλλά ίσως μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε αυτό το θέμα, τη συζήτηση. Κύριε Ρικέ, μιλάτε για το συντονισμό των περιβαλλοντικών πτυχών, πώς μπορούμε να τις ε, συνδυάσουμε με τις ε, μεταφορές της θαλάσσιες οδούς. Νομίζω ότι σε κάθε έργο και πρέπει να το να πούμε ότι το βλέπουμε και στον, στην περιοχή Ρήνου Δουναβή. Να δούμε πώς δηλαδή μπορεί να γίνει εφικτό αυτό το οποίο επιδιώκουμε. Και βέβαια πάντα πριν ξεκινήσει μελετάμε τις περιβαλλοντικές συνέπεια στον αντίκτυπο του περιβαλλοντικό. Είναι πολύ αυστηρή νομοθεσία. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς να τηρηθεί η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Και πάντα προσπαθούμε βεβαίως και αξίζει τον κόπο, είμαι πεπισμένη αν δεν ήμουν πεπισμένη ότι αξίζει τον κόπο, δεν θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά που κάνω. Πάντως, εάν μπορέσουμε να συγκεράσουμε τις δύο αυτές πτυχές, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι αν καταφέρουμε να τις συγκεράσουμε, λοιπόν. Θα πρέπει να επισημάνω το εξή, ότι, ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε την περιοχή του, του Δούναβη κατά τρόπο ολιστικό, διότι το, να ενισχύσουμε τις μεταφορές με τις θαλάσσιες οδούς αποσυμφορίζει τις χερσαίες οδούς. Και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε η προσπάθεια με την Ατζέντα 2020, γιατί τη φύση την επηρεάζουν και οι χερσαίες οδοί, όχι μόνο οι πλωτές οδοί. Τόσο οι χερσαίες όσο και οι σιδηροτροχές μπορούν να επηρεάσουν. το περιβάλλον. Μην κοιτάμε λοιπόν τα πράγματα με παροπίδες, ε, όπως το άλογο, αλλά κοιτάμε ολιστικά τη συνέπεια ενό προγραμμάτου. Έτσι λοιπόν, εάν μπορούμε να εξοικονομήσουμε, να περιορίσουμε τις ε, χερσαίες οδούς, αλλά και τις σιδηροτροχές, τότε νομίζω έχουμε καταφέρει πολλά. Θα καταφέρουμε πλήρως τα πολλά πιστεύω και για το περιβάλλον. Και θα δούμε ασφαλώς και την ανταπόδοση Για το ομόλογο έργο. Βεβαίω. Είναι μάλιστα έργο μεγάλης πνοής αυτό το οποίο συζητούμε και έστω και αν ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται τα ομόλογα έργου, θα έχει κάποιο νόημα να τα αξιοποιήσουμε. Και το ερώτημα βεβαίω είναι αν θα προλάβουμε εγκαίρως να τα χρησιμοποιήσουμε. έχουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ξέρετε, η δική μου εμπειρία από τη δική μου την περιοχή είναι ότι υπάρχουν τόσα διαθέσιμα κονδύλια, τέτοια λεφτά στον κόσμο. Φερρυπίν τα, τα Αυστραλιανά στα εξωτικά ταμεία που περισσεύουν και δεν έχουν τι να τα κάνουν τα λεφτά αυτά. Άρα το πρόβλημα δεν είναι τα λεφτά, λεφτά υπάρχουν. Πώς θα τα αξιοποιήσουμε είναι το πρόβλημα. Και πώς θα πείσουμε και τη γαλλική κυβέρνηση ότι είναι καλό το έργο, ότι μπορεί να φέρει και θέσει εργασία κτλ. Και πέραν τη Γαλλία, το Βέλγιο. Τα δύο Βέλγια, λέει η ομιλήτρια, η Βαλονία και η Φλάνδρα. Έχουν ήδη κάνει επενδύσεις, καθένα στη χώρα του, προσβλέποντας σε αυτά τα έργα. Θα ήταν κρίμα λοιπόν να μην προωθηθούν τα έργα. Το δε έτος 2003 με επίτροπο την κυρία Ντεπαλάσιο Ήμουν ε, υπουργό και υπογράψαμε σχέδια έργων που θεωρούσαμε μαζί με τη Γαλλία ότι είναι πολύ σημαντικά και τα στείλαμε προς έγκριση του Συμβούλου που ήταν εκνομόφωνα. Ήταν πολύ μεγάλη σημασία. Ήδη τότε. Αλλά από την άλλη μπορεί η κυβέρνηση της Γαλλίας να αντιμετωπίζει κάποιες οικονομικές δυσκολίες από ό,τι λέγεται. Να, δύο λεπτά μου είχατε δώσει. Καλά. Λοιπόν, τότε η κρίση Βεβαίω θα επηρεάσει τι εξελίξει. αναλόγως και τις απαντήσεις και τις θέσεις των κρατών όπως της Φλάνδρας και της Βαλονίας. Τι άλλο μου είχατε πει? Η κυρία Μέις Για το αν θα έχουμε τίποτα έτοιμο πριν το 2030. Όχι, βασικά είναι μακροπρόθεσμα σχέδια αυτά. Και χαίρομαι που είναι διατεθειμένες η Βουλγαρία και η Ρουμανία να αναλάβουν από κοινού την, ε, την κατασκευή ε, για το κομμάτι που αφορά τις χώρες και τον Δούναβη. Πρόκειται για ένα θαύμα συνεργασίας ασφαλώς, ε, μεγάλο έργο. Κύριε Κράμερ, λέτε ότι έχουμε 20% λιγότερο. Αλλά αν δεν κάνουμε τίποτα σε μερικά χρόνια θα έχουμε ακόμα λιγότερα. Διότι αξιοπιστία δεν υπάρχει επιχείρηση που θα επενδύσει σε σκάφη αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ποταμό δεν θα υπάρξει καμιά επένδυση. Και άρα δεν θα έχουμε και μεταφορές δράσεις, μεταφορές στο Δούναμι. Εάν προκύψει ξηρασία και κατέβουν τα επίπεδα των υδάτων στον ποταμό, δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει κανένα πλοίο. Και άρα ποιος θα πάει να επενδύσει σε πλοία όταν δεν είναι σίγουρος ότι ανά πάσα εποχή του χρόνου μπορεί να μεταφέρει, να κάνει τις μεταφορές του κατά τρόπον ε, ε οικονομικά συμφέροντα. Αυτό δεν κάνουν επιχειρήσεις. Εάν ξέρουν ότι μπορούν να στηριχθούν στην πλευσιμότητα του ποταμού, τότε θα το κάνουν. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κατάσταση ως ε, ε, αποδεικτικό για το δικό σας επιχείρημα, ως στήριγμα για το δικό σας επιχείρημα. Αντιθέτως αποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει κάτι. Όσο δεν γίνεται τίποτα η κατάσταση είναι αυτή που θα έχουμε. Τι να σας πω, να είχαμε πιο πολύ νερό. Μα αν δεν κάνουμε τίποτα, δεν θα μείνουν σκάφη στο νερό. Μετά μιλήσατε για τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Βαυαρίας που είχε ταχθεί κατά. Μπορεί, μπορεί. Αλλά εγώ ήμουν στο, στη βραδιά για τους κυριοβουλευτικούς στο Βερολίνο, για τους βουλευτές στο Βερολίνο, όπου υπήρχε εκπρόσωπο τη κυβέρνηση που τάχθηκε υπέρ. Άρα δεν ξέρω εάν η Βαβαρία ίδια ή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ταχθούν ε, αναφανδόν υπέρ του σχεδίου. Δεν είμαι και τόσο ισχυρή ώστε να πείσω τους πάντες. Θα δούμε τι θα γίνει στην ελεφαντομαχία που διαγράφεται. Ehm, Ο κ. Φαντάλε, ανάλυση κόστους αποτελέσματος πολύ θετική, έγινε. για το τι προκύπτει από ένα μεγάλο έργο. Ξέρετε ότι έχουμε στην Ολλανδία τέτοια εμπειρία. Από τη μια βάζουμε το κόστος, από την άλλη πλευρά της πλάστικας το, το, κέρδος, τα ωφέλη. Και βλέπουμε τι μπορεί να προκύψει σαν ισορροπία. Ιδάλλως. Εάν δεν είναι θετική ο απολογισμό, δεν γίνεται το έργο. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα. Εάν προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε πιο οικολογικά πλοία με νέες κινητήρες και πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και στις αγορές. Έχει δίκιο ο κύριος Κράμας. Πρέπει να πείσουμε και τους μεταφορείς των χερσαίων μεταφορών ότι μπορούν και πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στις πλωτές οδούς. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το αν θα φτάσει κάτι εγκαίρος πάντοτε. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά, αρκετά εμπορεύματα που δεν είναι νοπα λαχανικά που πρέπει να φτάσουν την άλλη μέρα το πρωί σε κάποια αγορά για να πουληθούν. Υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι τόσο ε, αναλώσιμο. δεν χαλάνε τόσο εύκολα. Ναι. Πολύ σύντομα να ολοκληρώσω. Με παραξενεύει λίγο το ερώτημά σας, γιατί υπάρχει ομάδα monitoring, ομάδα παρακολούθησης, που είναι γνωστή, ειδική του περιβάλλοντος, και όταν έρθει η ώρα για την εκθεσή τους, που δεν ξέρουμε αν θα είναι θετική ή αρνητική, αν θα έχει θετικό ή αρνητικό πόρισμα, σε τρεις μήνες περίπου πάντως, κάπου το Μάρτιο, θα γίνει η αξιολόγηση του αν πρέπει να προχωρήσουμε έτσι ή όχι. Και έτσι θα έχουμε στη θέση μας όλες τις πληροφορίες που πιστεύω κάθε ομάδα οικολόγων μπορεί να μελετήσει. Υπάρχει όμως η ομάδα του monitoring, η ομάδα παρακολούθησης ειδικά για αυτό το σκοπό. Ακούστηκε μια αντίρρηση για τον Ρήνο Μάιν και Δούναβη. Για το συνδυασμό, όχι για τη δουλειά που γίνεται. Ο Ματσιού Γκρούς ρώτησε για τις στενοπούς, τις νέες στενοπούς που τις ε, προβλέπουμε. Αυτό το ρώτησε και ο κύριος Κράμερ. που ζήτησε εξαίρεση για την κατηγορία 4. Ναι, κύριε Κράμερ, μπορεί να γίνει παντού εξαίρεση. Μόνο που δεν θα το πληρώσουμε. Εξαίρεση μπορεί να γίνει. Θέλετε να επιβάλλετε εξαίρεση για ολόκληρο το Δούναβι, κανένα πρόβλημα. Αλλά από την Ευρώπη δεν θα μπουν λεφτά σε αυτή την προσπάθεια. Ολόκληρο το Δούναβι μπορείτε να υπαγάγεται στην κατηγορία 4. Εάν όμω θέλετε να αξιοποιήσετε τι δυνατότητε αυτέ για τι επιχειρήσει τον τρόπο ωφέλιμο και οικονομικό, τότε πρέπει να γίνει διαφορετικά. Και οι στενοποιοί, εάν είναι υπερβολικέ, όπω βλέπουμε τώρα δυστυχώ να γίνεται στην Ουγγαρία, γιατί η Ουγγρική κυβέρνηση δεν συνεργάζεται, α το πω έτσι. ενδέχεται να προξενήσει σχολής, γιατί μπορεί να φτάσουμε να έχουμε όλο τον ε, Δούναβη όπως τον θέλουμε και να αποσύρει το κομμάτι της Ουκαρίας. Πάντως δεν είναι πια δίκτυα ευρωπαϊκά, είναι πραγματικά διευρωπαϊκά δίκτυα. Είναι καταπληκτική δουλειά. Και ακόμα μια λέξη, γιατί θα πρέπει σε μερικά λεπτά να αποχωρήσω. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου ευγενικό, αλλά κάνει μια αποχαιρετιστήρια δεξίως ο υπουργό και ήθελα να τον αποχαιρετήσω ειδικά αυτόν που ήταν υπεύθυνο και έχει κάνει πολλά πράγματα για την ε, Ζηλανδία στην περιοχή μου. Βεβαίως, λέει ο κύριος ε, Σίμψον, Σα ευχαριστούμε πολύ και δείχνουμε κάθε κατανόηση. Έχουμε κάπως καθυστερήσει προς το πρόγραμμα μας, δεν φταίτε μόνο εσείς, αλλά και εγώ. Καλωσορίζω εκπροσώπους της περιοχής Πολκαπάκη της Πολωνίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα παρακολουθήσουν την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών και τώρα παρακαλώ το τον κύριο Βίνκ να λάβει το λόγο για πολύ περιορισμένο χρόνο, 10 λεπτά μόλις. Έχετε το λόγο εσείς. Για το ERT εμείς. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 2012 ήταν πολύ δραστήρια τα πράγματα και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίως μας οδήγησε σε καλά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα στους σιδηροδρόμους. Το 2012 τι συνέβη. Καταρχάς ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τεχνικές προδιαγραφές ε, για τις μεταφορές πολλαπλών μέσων και 16 Απριλίου του 2012 υπεγράφηκε το Μνημόνιο Συνεννόηση στην Κοπεχάγη, ε, ημερομηνία που ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας, διότι Καταρχάς διευκρίνησε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μέσω των προθεσμών που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το ERTMS ε, θα είναι πλήρως συμβατές στις σιδηροδρομικές γραμμές και θα επανέλθω σε αυτό ιδίως όσον αφορά τις ημερομηνίε. Κατόπιν είχαμε την ε, τεχνική ολοκλήρωση και τη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων που παραδίδονται από διάφορους προμηθευτές και το σημαντικό στοιχείο εδώ ήταν οι δοκιμές. Και επίσης ε, αποφασίστηκε ότι πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικοί σιδηρόδρομοι όσον αφορά τις μεταφορές, γι' αυτό ακριβώ και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο μνημόνιο για τη μείωση του κόστους. Η μείωση του κόστους δεν αφορά μόνο το λογισμικό και το hardware ενός συστήματος, αλλά είναι και θέμα μηχανικής το να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε τα συστήματα και τις υποδομές σε τοπικό επίπεδο και επίσης να εναρμονίσουμε τις διάφορες διαδικασίες ε, έγκρισης και διοδότησης που υπάρχουν στην Ευρώπη, διότι υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος ε, και ε, απώλεια χρόνου και απώλεια χρημάτων. Το σημαντικό επίσης, το οποίο συνέβη επίσης στις 16 Απριλίου του 2012, ήταν ότι υπεγράφησαν και οι συστάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για την ε, βασική γραμμή 3. Θα θυμάστε ότι το 2008 αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μια βασική γραμμή γραμμή η οποία θα εγγυάται τη διαλειτουργικότητα, αλλά υπήρχαν και αρκετά σημεία και αρκετέ λειτουργίε, οι οποίε δεν υπήρχαν σε αρκετά κράτη-μέλη, κυρίως στη Γερμανία. Και έτσι το 2008 αναλάβαμε τη δέσμευση να καθορίσουμε και να αναπτύξουμε μια βασική γραμμή 3, μια baseline 3 που θα περιλαμβάνει και αυτή την επιπλέον λειτουργία. Και ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο είναι ότι το 2008 αναλάβαμε τη δέσμευση να ολοκληρώσουμε όλο αυτό μέχρι το 2012 και χαίρομαι ιδιαίτερα και είμαι περήφανο που όλοι διαφορεμονή. Ο οργανισμός, ε, το δίκτυο των διευρωπαϊκών δικτύων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκαν να έχουμε αποτελέσματα το 2012 και τα καταφέραμε και αυτό επιτύχαμε στις 16 Απριλίου του 2012. Τώρα την έχουμε λοιπόν αυτή τη γραμμή 3 και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να υλοποιήσουμε τη διαλειτουργικότητα. Αυξάνεται επίσης και η αξιοπιστία των δεσμεύσεών μας και πρέπει να σας πω ότι κάποια από τα κράτη-μέλη είναι πλέον θετικά διατίμων κείμενοι ως προς την ανάπτυξη αυτού του ευρωπαϊκού ε, συστήματος διαχείρισης των σιδηροδρομικών ε, διαδρόμων. Επίσης είναι πολύ σημαντική διότι μας παρέχει ευελιξία ε, και ως προς τις υποδομές αλλά μας παρέχει και μεγάλη ευελιξία ως προς το τοπικό δίκτυο και επέμενα ευθύ εξ αρχής ε, το λέγαμε ότι οι υποδομές μπορεί να είναι δύο 030 ε, ή ε, η βασική γραμμή 3 δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ γιατί υπάρχει συμβατότητα. Αλλά τα τοπικά δίκτυα θα πρέπει να έχουν τη βασική γραμμή 3 διότι αυτό μπορεί να δουλεύει και στο 230D και στη βασική ε, γραμμή. Επομένως μας παρέχει ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό φυσικά μπορούμε να το εγγυηθούμε και στην baseline 3 η οποία ε, παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2012. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το μεγαλύτερό μας επίτευγμα, αυτό που προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί, ώστε να το επιτύχουμε εντό του 2012. Τώρα, τι περιμένουμε για το εγγύς μέλλον. Καταρχάς, υπάρχουν κάποιες χώρες κράτη-μέλη, οποία, οι οποίες αποφασίζουν πλέον ότι αλλάζουν εντελώς το σύστημα σηματοδότησης ε, και ελέγχου σε ERTMS. Η Δανία και η Ελβετία επίσης αποφάσισε. Επίσης η Αυστρία, το Βέλγιο και σύντομα οι κάτω χώρες, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν εντελώς το σύστημά τους και να ε, συμπεριλάβουν το ERTMS. Και αυτό επιβεβαιώνει ότι το ERTMS δεν είναι πλέον θέμα συζήτηση. Ε, το μόνο θέμα είναι πώ θα το εφαρμόσουμε και πώ μπορούμε να επιλύσουμε τι δυσκολίε που μπορεί να ε, υπάρξουν από την εφαρμογή του. Μια μεγάλη αλλαγή επίση είναι ότι η Γερμανία άλλαξε στάση. Υπό την έννοια ότι πλέον είναι διατεθειμένη από τον Απρίλιο του 2012 και τούδε, έκαναν και αρκετέ συνεδριάσεις με του εκπροσώπους τη ε, γερμανική κυβέρνηση και του αρμόδιου γερμανικού υπουργείου, αλλά και με την Deutsche Bahn και συζητήσαμε αρκετά ε, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ε, ERTMS και πλέον η γερμανική κυβέρνηση είναι πεπισμένη ότι υπάρχει κάποιο σημαντικό πλεονέκτημα στην αλλαγή σε ERTMS και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία ακόμα, είμαι βέβαιος ότι ε, και σε υπουργικό επίπεδο και σε επίπεδο γερμανικών σιδηροδρόμων, τουλάχιστον ο διάδρομος 1, που είναι ο βασικός διάδρομος μέχρι τη Γενέβη, τον οποίο εξετάσαμε με πάσα λεπτομέρεια, και τώρα εξετάζεται το σύστημα Baseline 3 για το ε, ERTMS ε, για να εφαρμοστεί εκεί. Αυτή τη στιγμή εφαρμοστεί στο διάδρομο 1 μπορούμε να αποδείξουμε από εκεί και πέρα και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα στους υπόλοιπους διαδρόμους και αυτό φυσικά ε, θα είναι θέμα ευρωπαϊκής ανάπτυξης από εκεί και πέρα. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σταθεροποιήσουμε το πρότυπο, διότι υπάρχει το πρότυπο, και θέλουμε και εμπειρία φυσικά από την εφαρμογή τους στους ε, διαδρόμους και πρέπει να επιλύσουμε και το πρόβλημα του ESMR. Στο ERTMS έχουμε την... το συνδυασμό του ETCS και του ATMS και πολλοί ενδιαφέρονται ε, για τις ε, παρεμβολές που μπορεί να υπάρχουν στα συστήματα GSM και γι' αυτό έγιναν και αρκετές επαφές και με τις ε, υπηρεσίες ε, επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών για να δούμε τι γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα. Τώρα, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά όλο αυτό, θα πρέπει αφενός να υποστηρίξουμε και την τεχνική πτυχή του ERTMS, αλλά φυσικά και όλες τις ε, ε, οδηγίες που αφορούν ε, τους ε, κανονισμούς και τους, την νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Τώρα, εάν το ERTMS θέλουμε να είναι επιτυχημένο, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι να υπάρχει συμβατότητα και μεταξύ των σιδηροδρομικών γραμμών, αλλά και του εξοπλισμού που υπάρχει επί του σειρμού, γιατί θα πρέπει όλα αυτά να είναι συμβατά. Το κόστος επιμένω ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, θα πρέπει να υπάρχει baseline 3 για να υπάρχει ευελιξία. Επίσης, εξοπλισμό των διαδρόμων βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξης ε, μέχρι το 2020. Είμαι αρκετά ρεαλιστής και γνωρίζω ότι σε κάποια κράτη-μέλη θα δημιουργήσει πρόβλημα η τήρηση της προθεσμίας, αλλά εμείς αναμένουμε οι αλλαγές ε, που πρέπει να γίνουν για κάθε διάδρομο σε κάθε κράτος μέλος να μας δοθούν μέχρι το τέλος του έτους και αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά, θα απαντήσουμε για να δούμε τι μπορούμε να υλοποιήσουμε σε ρεαλιστικά πλαίσια. Ε, υπάρχουν κυρίως ε, χρηματοοικονομικοί περιορισμοί για, την, ε, για τις επενδύσεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση του τοπικού πληθυσμού και αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα πρέπει να εξορθολογήσουμε την ε, εθνική διαδικασία έγκρισης με, στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα τη μείωση του κόστους, αναφερθήκαμε στις οικονομικές ε, πτυχές για τις πλωτές οδός, αλλά νομίζω ότι και για τους σιδηροδρόμους θα πρέπει να συνειδητοποιούμε πάρα πολύ καλά και ποια επιχειρησιακά σχέδια θα πρέπει να συνδέουμε με όλα αυτά και θα πρέπει να πιέζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και κατόπιν, την εφαρμογή των διαδρόμων μεταφοράς εμπειροφμάτων. Εδώ ε, να σας διαβεβαιώσω, εξότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, ότι είμαστε οργανωμένοι αρκετά καλά για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Υπάρχει οργάνωση και για λειτουργία των ε, διαδρόμων ε, και τα εκτελεστικά συμβούλια και τα αρμόδια υπουργεία που ασχολούνται με αυτά. Για να λειτουργήσει και να υλοποιηθεί το business plan. Αλλά σε επίπεδο επιτροπής έχουμε επίσης και τα δύο επίπεδα για την παρακολούθηση με την ε, Διευθυντική Επιτροπή που παρακολουθεί και τα θέματα του RTMS και την ομάδα που παρακολουθεί την υλοποίηση όχι μόνο του RTMS αλλά και του κανονισμού ε, για του σιδηροδρόμους. Άρα σε δύο επίπεδα γίνεται η παρακολούθηση. Τι θα πρέπει να κάνουμε τους προσεχείς μήνες και το 2013. Όσον αφορά τα μέσα που έχουμε στη θέση μας, μπορούμε πιστεύουμε να αξιοποιήσουμε τις επενδύσεις ε, που προβλέπονται ε, μπορώ να είμαι ικανοποιημένο ότι είχαμε στήσει 500 εκατομμύρια το 2007 και μπορέσαμε να τα διατηρήσουμε με επιπλέον 100 εκατομμύρια σε μια πρόσκληση που είχαμε εκδώσει και άλλη μια τώρα που θα μας φέρει άλλα 100. Βέβαια περιμένουμε περισσότερες επενδύσεις γιατί και οι επενδύσεις ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Και εν όλο, αν κοιτάξουμε τι επενδύσεις γίνονται για το ERTMS, είναι περίπου 1,2-1,3 δις περιφέρειες και διευρωπαϊκά μαζί. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε το ERTMS, να αποφύγουμε, και αυτό είναι το πρόβλημα και η παγίδα της καθαρά εθνικές επιλογές, το προσανατολισμό των εθνικών. Να αξιοποιήσουμε στο δυνατόν τυποποιημένο εξοπλισμό η RTMS, που θα μειώσει και τις τιμές, και να περάσουμε στο Base 93. Για τους σιδηροδρόμους και τους σιδηροδρόμους έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με το υλικό και το, το ανθρώπινο και το τεχνικό που έχουμε, με τρόπο συστηματικό, να έχουμε καλύτερη ορατότητα στις υποδομές, να λάβουμε υπόψη το σχετισμό μεταξύ διαδρόμων και τερματικών που αποτελούν και το σημείο επικοινωνίας των διαφόρων μέσων μεταφορός και να δώσουμε πρόσβαση ελεύθερη στους διαδρόμους. Πριν όμως σταματήσω, πρέπει να φτάσω στα συμπεράσματά μου και πριν από αυτό θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα σύντημα το οποίο έχω να κάνω σχόλια. Θέλω να πω ότι το έχουμε συστήσει και με άλλου τονιστέ. Πρέπει να βελτιωθεί, να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ μα για του σιδηροδρόμου και το τι κάνουμε, τι προσφέρουμε στον ε, πολίτη, ιδιαίτερα δηλαδή η επικοινωνιακή πτυχή, να γνωρίζει κανείς τι γίνεται για τις κοινότητές μας. Δεν είναι αρκετά αυτά που γίνονται και δεν είναι πιστικά για τον πολίτη, τουλάχιστον όσον αφορά το σιδηρόδρομο ως μέσο μεταφοράς. Έχουμε βεβαίως ως βάση το βασικό δίκτυο που έχει παρουσιαστεί και προταθεί στο Κοινοβούλιο. Κλείνω λοιπόν. Έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ηγεσία, ηγετική θέση προς την τεχνογνωσία, την τεχνολογία. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα από την βιομηχανία ως προς το ERTMS. Και δεύτερον, και μια από τις κύριες προτεραιότητες, τώρα ανέλαβα τη θέση του συντονιστή, ε, προχωρούμε και φτάνουμε στο σημείο άνευ επιστροφής και μπορώ να σας πω για πρώτη φορά στη ζωή μου ότι φτάσαμε τώρα στο σημείο άνευ επιστροφής. Το σύστημα ERTMS είναι το καταξοχήν μέσον και σύστημα για την Ευρώπη στο μέλλον. Ευχαριστώ. Γκρός και άλλοι. Από δύο λεπτά. Για να προσπαθήσουμε να δώσουμε λίγη τάξη στη συζήτηση. Ο κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Βίνκ. Κινείστε σε έναν χώρο που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι δεν είναι εύκολο. Και το χειρότερο είναι ότι οι περισσότεροι, οι πάντες, είναι πεπισμένοι ότι πρέπει να εργαστούμε κατά τρόπο στονισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο που ο άμεσος χρήστης, εκείνος που θα υποφεληθεί ευθέως από τον συντονισμό αυτών και τις ευρωπαϊκές προσπάθειες, δεν είναι πεπισμένος. Το Κοινοβούλιο λοιπόν, η, η Ένωση δεν έχει μάλλον κάνει καλή επικοινωνιακή πολιτική ως προς τα πλέον εκτήματα ενός στερεοδρομικού συστήματος για τις μεταφορές και φαίνεται ότι δεν έχουν επιστεί τα κράτη για τα πλέον εκτήματα των σιδηροδρόμων. Οι θα είχαν συμπεριφερθεί διαφορετικά. Δεύτερον, χρηματοδότηση. Και ρωτώ, γιατί ακούμε από διάφορες χώρες, αλλά ασφαλώς από το Βέλγιο μπορώ να το βεβαιώσω, κύριε Βίνκο, ότι έχουν περικοπεί σημαντικά οι προπολογισμοί για τα θέματα των σιδηροδρόμων. Θα λέγω ότι έχουμε φτάσει σε ένα ελάχιστο διαβίωσης ως προς τις σχετικές, τα σχετικά κονδύλια, που φέρει σε αμφιβολία ακόμη και την ασφάλεια των δικτύων. Επερωτώ λοιπόν στα άλλα κράτη τι εικόνα έχουμε τι συνέπειε μπορεί να έχει για τις μεταφορές και τι είδου επενδύσεις χρειάζομαι για να μην έχουμε τέτοιες ριζικέ περικοπές. Και τέλος, τεχνολογία. Μιλήσατε για το μνημόνιο συνεννόηση τη Κοπενχάγης. Βεβαίω και θα προτιμούσα να το είχαν υπογράψει όλα τα κράτη και οι υπουργοί, όχι μόνο επιχειρήσει. Μια και αναφερθήκατε και στη Γερμανία, που χαράζει το δρόμο στα θέματα αυτά θα πω ότι υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι εταίροι που δεν έχουν προσυπογράψει αυτό το μνημόνιο. Βλέπετε λοιπόν κάποια ευκαιρία, πιθανότητα, ε, δυνατότητα να διευρυνθεί η συμμετοχή, γιατί έχουμε και τη συζήτηση την επόμενη, στην οποία θα πρέπει να στηριχθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σολκαντράουι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, τον κύριο Βίνκ. Αισιόδοξο σας βρίσκω. Πολύ καλό αυτό. Για τη Γερμανία θα ήθελα να πω ότι είναι πολλέ οι επικρίσει που και εμεί είχαμε διατυπώσει βάρο Γερμανία και ίσω τώρα μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποια θετική εξέλιξη. Άρα ο συντονιστή έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Για τα προσεχή χρόνια τουλάχιστον ε, μπορεί να επηρεάσει τι εξελίξει και καλό θα είναι να προσπαθούμε να πείθουμε όσου μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτών των ε, έργων. Ερωτώ λοιπόν, ε, βλέπουμε μεγάλες προκλήσεις προς τη RTMS για το τροχαίο υλικό. Ε, ε, είναι όμως τόσο διαδεδομένη, έχει τόσο πολύ προχωρήσει η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στο τροχαίο υλικό, είναι εξοπλισμένο όλα τα τρένα. Μετά μας λέτε ότι ίσως να μην έχει προχωρήσει αρκετά η επεξεργασία του ERTMS, πολλά είναι τα διοικητικά προβλήματα ανάλογα με το κράτος μέλος, ξέρω ότι δεν είναι δική σας απαραίτητα αρμοδιότητα, αλλά... Πρέπει να κάνω την ερώτηση, μια και θα γίνει η συζήτηση για την ε, υπηρεσία σιδηροδρόμων της Ευρώπης. Τι είδου αρμοδιότητες εσείς θα λέγατε ότι πρέπει να περάσουν από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία σιδηροδρόμων, για να λειτουργούν καλύτερα τα δίκτυα. Και πού μπορείτε να εντοπίσετε τις δυνατότητες για ε, οικονομία κλίμακας, ε, ανάλογα με τα σχέδια, ανάλογα με την επικέντρωση των προσπαθειών κτλ. Κυρία Μάστινα, παρακαλώ δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση κύριε Ξέρουμε ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη και τονίστηκε από του προλαλήσαντε. Θέλουμε ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο όπου μπορεί κανεί να μπορεί να κυκλοφορεί αποτελεσματικά και τεχνολογικά να είναι εξοπλισμένο. Έρχομαι από τη Γερμανία και δεν είναι τόσο δίσκαμπτη, άκαμπτη η Γερμανία όπω πέρσι, αλλά δεν έχουμε τίποτα υπογράψει. Πώ πιστεύετε ότι θα προσυπογραφούν κάποια πράγματα για να σημειωθεί πρόοδο, διότι έχει άλλο σύστημα με άλλη τεχνολογία η Γερμανία σε σχέση με τη διαλυτική στην Ευρώπη, ίσως αυτό θα έθετε κάποια προβλήματα. Άλλη ερώτηση. Άλλες χώρες ε, δημιουργούν προβλήματα διότι είπατε ότι για το ε, διαδίκτυο αυτό είπατε ότι πολλές κυβερνήσεις είναι πεισμένες ότι πρέπει να γίνει αυτό, αργότερα όμως αναφέρθηκε ότι η επικοινωνία πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω και πρέπει να πιστούν οι άνθρωποι. Ποιοι πρέπει να πιστούν και πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε για να πείσουμε κάποιους. Το τελευταίο, αναφέρατε ότι εθνικές επιλογές θα πρέπει να αποφεύγονται. Ε, αναφέρεστε στη Γερμανία σε κάποιους άλλους που πρέπει να προσέξουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κράμερ δύο λεπτά παρακαλώ. Από την Κάρλα Πέρις έμαθα ότι αυτό δεν ε, δημιουργούσε πρόβλημα ναι. και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ για αυτά τα οποία κάνατε και μας είπατε. Τώρα, για το πώς ε, βρίσκονται κάποια πράγματα τα οποία ε, ίσως μπορεί κάποια προβλήματα να δημιουργούσαν. Εσείς ε, επανειλημμένα τοποθετηθήκατε. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις, τώρα πρόκειται για έναν διάδρομο. Χαίρομαι για το ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε και εκείνη να προχωρήσει. Έχει υπογράψει, θα υπάρξει προαγωγή. Χαιρόμαστε αν μπορεί να γίνει αυτό σε ένα διάδρομο. Όμως το ερώτημα παραμένει. Ποιος συντονίζει όλα αυτά τα πράγματα και θα μπορέσουν όλα αυτά να λειτουργήσουν ώστε για παράδειγμα εσείς θα καθορίσετε τι θα γίνει σε σχέση με αυτά τα θέματα για το σιδηρόδρομο ή θα περάσουν στα συναρμοδιότητα των κρατών μελών. Το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό. Και σε σχέση με, με το διαδίκτυο αν οι χώρες θέλουν τα δικά τους συμφέροντα και τις ιδιομορφίες να εντάξουν, αυτά δεν θα, είναι, ε, δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρέπει προς τα πάνω και προς τα κάτω να είναι σύμβατα και συνεκτικά όλα αυτά. Και η βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο να μην κοιτάζει μόνο τα συμφέροντά της και όχι την πρόσθετη ευρωπαϊκή αξία. Δεν είναι δυνατόν ε, να έχουμε ξεχωριστές ε, ε, κινητήριες μηχανές που θα πρέπει κάθε τόσο να αλλάζουν. Τι γίνεται σε σχέση με το πρόβλημα των τηλεφωνικών γραμμών. Έχει επανορθωθεί αυτό γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση, δεν υπάρχει όμως ακόμα η ευρωπαϊκή λύση. Ευχαριστώ. Κάντσιαν παρακαλώ, δύο λεπτά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον ε, συντονιστή, τον κύριο Βίνκ. Πολύ αισιόδοξο το έργο σας, ε, πολύ καλή η δουλειά σας μέχρι τούδε. Δύο ερωτήσεις να σας θέσω. Καταρχάς, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία εξετάζουμε στα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα, δεν προβλέπουν συντονιστή για το ERTMS και ε, λογικά θα κατανεμηθεί το έργο του στους 10 συντονιστές των 10 διαδρόμων. Το ερώτημά μου είναι, το εξής. Ε, είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας αυτός για τις μελλοντικέ εργασίες. Και αν όλες αυτές οι δικές σας αρμοδιότητες ε, κατανεμηθούν στις 10 διαδρόμους και απορρομηθούν εκεί, θα, θα έχουμε αποτέλεσμα κατά την άποψή σας, γιατί αυτό το χρειαζόμαστε στις επόμενες μέρες. Δεύτερον, στην έκθεσή σας αναφέρεστε ε, στην υποστήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρχει εναρμόνιση και τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ακριβώς για να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι διαλειτουργικό και θα είναι και λιγότερο γραφειοκρατικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαρτού για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φίνκ και για την παρουσίαση, για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ καλή. Μια ερώτηση. Δύο είχα βασικά, αλλά με κάλυψε ο κύριο Κάντσεν για την άλλη, για τη μία. Ε, ρωτώ λοιπόν για τις, ε, και σε σχέση με τη Γερμανία συγκεκριμένα. Γιατί είχα πρόσφατα μια πολύ φορτισμένη συζήτηση με τον εκπρόσωπο των γερμανικών συντηροδρόμων, όπου εν τέλει τον ρώτησα γιατί καθυστερεί εν τέλει τόσο πολύ η, εφαρμογή του, η εισαγωγή του ERT μας. Ε, μας είπε λοιπόν ότι το πρόβλημα ήταν και τεχνικά, η τεχνική ασφάλεια αλλά και η ασφάλεια των δεδομένων. Ρωτώ λοιπόν τι είδους μέσα μπορείτε να προσφέρετε, τι είδους δυνατότητες μπορούμε να έχουμε ώστε να προχωρήσουν αυτά τα, τα σχέδια πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να δώσετε σύντομα όσο το δυνατόν τις απαντήσεις σας, παρακαλώ κύριε Βίνκ. Πρώτα απ' όλα. Για την ερώτηση του κύριου Γκρός. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Επιμένω ότι ό,τι έχουμε καταφέρει στο παρελθόν, ό,τι έχει γίνει στην προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο, όπου είχαμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα τις επενδύσεις του μας κατά 50% του, του κόστους, πρέπει να επαναληφθεί, πρέπει να διατηρηθεί ως δυνατότητα και όχι μόνο για τις υποδομές, αλλά και για το υλικό πάνω στο τρένα, γιατί χρειάζεται αυτό το κίνητρο για τον χειριστή operator, για την εταιρεία μάλλον operator, ώστε να προχωρήσει. Αν δεν το έχει αυτό σαν κίνητρο, δεν θα το υλοποιήσει από μόνη της. Δεύτερον, θα πρέπει κίνητρα να δώσουμε επίσης για να περάσουν στο baseline 3 που προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία. Και θα έχουμε φαντάζομαι και άλλη ευκαιρία να πείσουμε τα κράτη-μέλη. Αλλά νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο πολύ να πείσουμε ότι να υπάρχει ένα σύστημα και πρέπει να το εξυπήσουμε, αλλά ότι ακόμα κοιτάνε τι κάνει η Γερμανία και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η Γερμανία με τέσσερις διαδρόμους που τη διασχίζουν. Και άρα, εάν η Γερμανία πάρει ε, την απόφαση να ενσωματώσει το ERTMS, να δεχθεί το ERTMS, τότε θα αποτελέσει αυτό και μόνος κίνητρο για τις άλλες χώρες. Ήδη νομίζω έχει σημασία αυτό και ως ε, πρόγραμμα επικοινωνιακό, νομίζω πρέπει να το κοιτάξουμε. Μια και μιλάμε λοιπόν για τη Γερμανία, θα έλεγα ότι μπορώ να είμαι αισιόδοξο, γιατί είναι και ο μόνο τρόπο να επιβιώσουμε και να προχωρήσουμε. Να επιβιώσει και να, και να προχωρήσει, αλλά διαβλέπω και μια αλλαγή στάσει και νοοτροπία. Μπορεί να μην μπορώ να μιλήσω με τον Υπουργό και το Υπουργείο. Ελπίζω ωστόσο, τουλάχιστον για τον ε, πρώτο διάδρομο, ότι μέσα σε μέρες, όχι εβδομάδες ή μήνες, μέσα σε μέρες θα μπορέσουμε να λάβουμε γραπτή συμφωνία για το ERTMS για το διαδρομό 1. Άπαξ λοιπόν και εξασφαλίσουμε τον διαδρομό 1, τότε ξεκινάμε τη συζήτηση και για τους άλλους και μέχρι το τέλος του 2013 μπορώ να ελπίζω, πρώτον Θεός, ότι θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε εδώ και να σας δώσω καλύτερες ειδήσει για τους λοιπούς διαδρόμους. Και μέσα βέβαια να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Επίσης πολλές διαφορές καταγράφονται ακόμη μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών λόγω της απαρχαιωμένης ε, νομοθεσίας ε, και της παλαιάς νομοθεσίας αν θέλετε, δηλαδή το να εγκαταλείψουν την εθνική νομοθεσία και να περάσουν στην ευρωπαϊκή πάντα αποτελεί μια δύσκολη μετάβαση. Ωστόσο υπάρχει δέσμευση. Το ERTMS το 2012 ήταν έτοιμο. Το κάναμε εμείς. Άρα λοιπόν υπάρχει η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το ψυχολογικό του είπε, επιχείρημα για να πείσουμε τους εταίρους. Βεβαίω, έχουμε την Επιτροπή Κινδύνου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορεί να συνομιλεί με τους εκπροσώπους των κρατών μελών για να του πείθει σε αυτό το επίπεδο. Άρα συνεχίζεται Συνεχίζονται οι επίεσει, συνεχίζεται η επικοινωνία, η επαφή για να πείσουμε και τα κράτη-μέλη και όταν βλέπουμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη περνάνε, ε, κάνουν πλήρη μετάφαση του ERTMS, πιστεύουμε ότι αυτά θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πάντως πρόκειται για μια από τις προτεραιότητες που έχουμε για να περιορίσουμε και το κόστος στην απώλεια χρόνου αλλά και χρήματος. Φαντάζομαι ότι αυτό καλύπτει και τις διατυπώσεις, γιατί τις οικονομίες κλίμακας ναι, Υπάρχουν τέτοιε δυνατότητε, εφόσον όμω είναι τυποποιημένο ο εξοπλισμό. Και εφόσον οι χώρε, τα κράτη-μέλη ή οι επιχειρήσει, ε, είτε για την ε, χορήγηση ε, του υλικού, είτε για τη διαχείριση, συμφωνήσουν και συμμετάσχουν σε αυτές τις οικονομίες. Για τις άλλες χώρες, κύριε Βάσνερ, άπαξ και υπάρξει συμφωνία, όπως είπα, της Γερμανίας, δίνει όθηση αυτομάτως και επικοινωνιακή και ουσιαστική στη συμμετοχή των κρατών, των λοιπόν κρατών. Ξέρουμε ότι ορισμένα κράτη θα διστάσουν, αλλά πάντα έχουν ένα μάτι στραμμένο στη Γερμανία όλοι. Η Γερμανία είναι και στο κέντρο της Ευρώπης τέλο πάντων και μετράει πάρα πολύ η δική της επιλογή. Άρα προσπαθούμε να πείσουμε και τις εθνικές υπηρεσίες βεβαίως. Και αν το καταφέρουμε αυτό, εν μέρη θα οφείλεται στην αλλαγή νοοτροπίας που ήδη σημειώνεται. Για τον κύριο Κράμερ. Οι έξι διάδρομοι. Ας ξεκινήσουμε τον πρώτο και μετά να δούμε και από την εμπειρία που θα έχουμε συλλέξει για να πείσουμε για τους λοιπούς διαδρόμους. Πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας μέσα σε μια διαρκή διαδικασία επικοινωνίας, επαφών με τα Υπουργεία, με τις αρχές, βιομηχανία. Λέτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για τα 600 χιλιόμετρα ακόμα. Ναι, αλλά αυτός είναι και ο στόχος. Δηλαδή το ERTMS, βασική γραμμή 3, στον διάδρομο 3, μπορεί να εγκατασταθεί στο διάδρομο 1. Και αυτός είναι ο στόχος, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε ένα τρένο από το Ρότερνταμ στη Γένοβα της Ιταλίας χωρίς διακοπή. λύσεις για τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά είναι ακριβές. Και άρα πριν να κοιτάξουμε τεχνικές λύσεις, πιο σημαντικό είναι να δούμε τι είδους συμφωνία μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις ε, επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιών, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των παρεμβολών που αναφέρατε. Επίσης, ε, για τον συντονιστή, η ορτή μας, προσωπική γνώμη θα σας δώσω, και θα αποφασίσετε βεβαίω εσεί ο ίδιο και η Επιτροπή ολόκληρη. Αλλά στο στάδιο αυτό, για να εξασφαλιστεί η τεχνική παρακολούθηση, συνέχιση τη εφαρμογή του ERTMS, θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται συντονιστή ERTMS για άλλα 7 χρόνια, αλλά τουλάχιστον για 2 χρόνια είναι απαραίτητο. Ή μη τι άλλο, μέχρι ότου εξασφαλίσουμε την υλοποίηση του πρώτου διαδρόμου. Απρόσκοπτη εφαρμογή και λειτουργία. Μέχρι τότε χρειάζεται αυτό ο συντονιστή. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι με τη δύναμη τη εμπειρία, τη γνώση και μπορούμε στη συνέχεια να διανοηθούμε την κατάργηση της θέσης του συντονιστή. Αλλά μέχρι τότε θα έλεγα τα δύο αυτά χρόνια επιπλέον, δύο ή τρία χρόνια να τα δώσουμε. Και για τον κύριο Ερτούκ, γιατί ήταν τόσο διστακτική, λέτε, για να, στην αποδοχή του ERTMS, η γερμανική στυρόδρομη. Νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν κυρίως χρηματοδότησης, όχι. Κύριος Κράμερ χωρίς μικρόφωνο. Ο κύριος Σίμψον χωρίς μικρόφωνο. έχουν προπολογισμούς ορισμένους για τις ε, επένδυσεις τους και ήταν δύσκολο να συμπεριλάβουν και τις πρόσθετες αυτές επενδύσεις στον, προ... στον ενιάυσιο τέλο πάντων προπολογισμό επενδύσεων και έπρεπε να συζητήσουν και με τα Υπουργεία, το αρμόδιο Υπουργείο το πώς θα γινόταν αυτή η επένδυση, πράγμα το οποίο κρατάει χρόνο βέβαια. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεολεβέρα τώρα για τους θαλάσσιους αυτοκινητόδρομους. Αν μπορέσετε να τηρήσετε και τα 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέχρι σήμερα έχουμε προχωρήσει και έχουμε 19 από αυτά τα προγράμματα που ήδη έχουν προχωρήσει και έχουν μια τελική επένδυση πάνω από έναν όγκο ενός δισεκατομμυρίου. Αυτά όλα τι καταδεικνύουν ότι ε, στο πλαίσιο αυτών των ε, οδών έχουμε μια ισχυρή πλατφόρμα για την υλοποίηση των τεχνολογικών προδιαγραφών για να βελτιωθεί η ποιότητα αυτών των ε, δράσεων και η ενσωμάτωσή τους μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταφορών. Να υπενθυμίσω κάτι εδώ, ότι έχουμε δέκα βελτιωμένες διασυνδέσεις, θαλάσσιες διασυνδέσεις ναυτιλιακές διασύνδεσεις σε σχέση με αυτά και εννέα ευρύτερου ωφέλους προγράμματα που τα αποτελέσματά τους θα διαχυθούν και θα διαδοθούν ευρύτερα. Η προαγωγή των αυτοκινητοδρόμων στη θάλασσα και η ανάπτυξη πολλών μικρών δράσεων που συνολικά έχουν βελτιώσει τους εξής κυριότερους άξονες ε, την πρόσβαση και την διασύνδεση λιμάνων, το, λιμένων, το σύστημα πληροφόρησης, την αποτελεσματικότητα των δράσεων και την βελτίωση υποδομών για τη διασύνδεση λιμένων. Όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο των ε, ε, ναυτιλιακών διασυνδέσεων οδήγησαν στο να προαχθούν καινοτόμε δράσει σε συνδυασμό με πρακτικές λύσεις, για παράδειγμα εφείς υποδομέ και τεχνολογίες ε, ε, LNG. Σε αυτές τις ε, περιπτώσεις είχαμε πιλωτικές δράσεις που αναπτύχθηκαν που αναμένουμε να δώσουν πρακτικά χειροπιαστά αποτελέσματα. Το να ενοποιήσουμε αντί να κατακαιρματίσουμε ήταν ο στόχος. Οι δραστηριότητες Motorways at Sea έχουν σημαντικό ρόλο. Προάγουν την ανάπτυξη λειτουργικών προδιαγραφών και διατάξεων και κοινών ε, λειτουργικών διατάξεων και βέλτιστων προδιαγραφών στο benchmarking. Εν συντομία, Motorways at Sea αντανακλούν απαιτήσει πολιτικών ώστε να μπορούν να εξευρεθούν οι βέλτιστες ευρωπαϊκές λύσεις στα προβλήματα. Η επιτυχία αυτή μπόρεσε να επιτευχθεί με την προώθηση της συνειδητοποίησης των εμπλεκόμενων για τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τις κοινέ δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν. Δημιουργείται μια βάση συνεργασίας μεταξύ λιμένων και περιοχών, θαλάσσιων περιοχών, όπως π.χ. της περιοχής της Βαλτικής. Μια κοινή κατανόηση των δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας καθώς επίσης ε, και προαγωγή των θεμάτων ασφάλειας ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί μέσα από αυτή τη συνεργασία να αναπτυχθούν αυτοί οι στόχοι βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Αδριατική, έχουμε και την συνεργασία διαφορετικών ε, λιμένων, π.χ. στο βορρά της Αδριατικής, ώστε να αντιμετωπιστούν ε, οι, τα κενά και οι αδυναμίες και να προαχθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων σε αυτές τις περιοχές ώστε να έχουμε και την περιοχή της Μεσογείου και της ε, Μαύρης Θάλασσας, ε, του Εύξηνου Πόντου και της ε, Βόρειας Όχθης της Αφρικής με την ευφυή δράση χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και εργαλεία ώστε να έχουμε ένα ευρύ φάσμα δράσεων ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί π.χ. για παράδειγμα με το Μάρκο Πόλο και με τις δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων με κάθε ένα εξειδικευμένο σε συγκεκριμένο πεδίο δράσεων. Γενικά οι υπηρεσίες Μάρκο Πόλο για τη χρηματοδότηση ενώ βλέπουμε ότι έχουμε και την, ε, τον, την εστίαση στις υποδομές και στα συστήματα πληροφόρησης, π.χ. επιμελητιακή υποστήριξη, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στοχεύουν στην ε, στη διάθεση 300 εκατομμυρίων για τις ε, λεωφόρους της θάλασσας ε, για τον προγραμματισμό 2007-2013 σε αυτή τη χρονική περίοδο. Για την περίοδο 2014-2020 αναμένεται η υποστήριξη ότι θα αυξηθεί σε επίπεδα που θα είναι επαρκέστερα για τις ανάγκες αυτές Γνωρίζετε ότι το εξωτερικό εμπόριο της Ευρώπης εξαρτάται πάνω από 70% από αυτού του είδους της δράσης και 40% σε σχέση με το εσωτερικό εμπόριο. Προτεραιότητες λοιπόν για το 2012 ε, είναι οι εξής, είναι οι εξής ακόλουθες η ομαλή ενσωμάτωση των διαδρόμων των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, διασύνδεση χερσαίων μεταφορών, παράθυρα ε, δυνατοτήτων διασύνδεσης και η δυνατότητα να υπάρχει ε, η αξιολόγηση αυτή που θα διασφαλιστεί μέχρι το 2015. Να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ε, που πρέπει να αντιμετωπιστούν LNG, ε, αναπλήρωση, ε, αναφόρτιση κτλ. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι οι ε, δυνατότητες ελέγχου από πλευράς περιοχών έχουν καθορίσει το μέγιστο όριο το οποίο μπορεί να, μπορεί να οδηγήσει στην έγκριση από τα κράτη-μέλη πρέπει να δούμε ότι έχουμε και την προσφορά ευκαιριών για την αγορά με νέα κτίρια, με την, τον εξοπλισμό, με την ε, ε, δυνατότητα ανεφοδιασμού και την ε, λήψη υπόψη της ναυπηγικής βιομηχανίας. Όλο και περισσότερο η ασφάλεια γενικά με την εκπόνηση διατάξεων ε, που πρέπει να προαγάγουμε στις βιομηχανικές μας δράσεις. Αναμένεται ότι οι νέες προτεραιότητες και εργαλεία που προτείνονται μέσα από αυτό το πλαίσιο που αναμένονται ότι θα ξεκινήσουν στις 28 Νοεμβρίου και ιδιαίτερα οι πιλωτικές δράσεις θα συνεχίσουν να ε, ενδιαφέρουν τους ε, εμπλεκόμενους στην αγορά. Αυτό το, μέλο, αυτό το εργαλείο θα δίνει τη δυνατότητα πλήρους δοκιμής χωρίς ε, να θίξουμε τα θέματα ανταγωνισμού. Θα δώσει τη δυνατότητα ολοκληρωμένα να ενταχθούν θέματα ε, λειτουργικότητας ε, με τη βελτίωση των δυνατοτήτων μεταφορών ώστε να ξεκινήσουν οι φάσεις εφαρμογής άμεσα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πιλωτικών δράσεων. Αυτό είναι ακριβώς η πεμπτουσία της ε, προσπάθειας για καινοτομία, καινοτόμο δράση παρέχοντας συνδρομή και υποστήριξη με αυτά τα υψηλής τεχνολογίας εργαλεία για την αύξηση, βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μεταφορών όπως π.χ. των αναγκών τελωνίων με ηλεκτρονική κατάθεση φορτωτικών και ε, εγγράφων που συνοδεύουν τα φορτία θα μπορέσουν να συνεισφέρουν όλες αυτές οι διεργασίες στο να διευκολυνθούν οι τελωνιακές διαδικασίες, διεργασίες και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα από την πλευρά των μεταφορών. Είναι ένα κλειδί για την ε, ευημερία και την πρόοδο στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε την ε, πραγματική αυτή προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί σε αυτού του είδους τις μεταφορές με τα αναγκαία κονδύλια. Υπενθυμίζω ότι το τρέχον χρηματοδοτικό πλαίσιο 2007 έως το 2013 έχει έναν όγκο περίπου 3,5% των συνολικών πόρων, δηλαδή περίπου 500 εκατομμύρια αυτού του είδους ε, τα ποσοστά, αυτού του είδους το ποσοστό είναι σαφώς ανεπαρκές για να μας οδηγήσει στο να αντιμετωπίσουμε τις συντριπτικές ανάγκες ε, που έχουμε για την επόμενη περίοδο που ε, πρέπει να καλυφθεί 2014-2020. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι θα απαιτηθούν πάρα πολλές προσπάθειες για να τα βγάλουμε πέρα αυτή, με αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. It's all minutes each. Από δύο λεπτά στον καθένα ούτως ή άλλως θα δώσω. Ο κύριος Καντσιάν, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τον κύριο Ντεολιβόηρα, εξαιρετική η αλλως θα δωσω ο κυριος καντσιαν για δυο λεπτα παρακαλω ευχαριστω τον κυριο ντεολιβοηρα εξαιρετικη δουλεια σας. Νομίζω ότι η θαλάσσιοι αυτοκινητόδρομοι είναι θεμελιώδους σημασίας. αποδοτησουμε τις αγορές μας Θεωρώ όμως ότι μία πιο αποφασιστική ε, δράση για να αναπτύξουμε προγράμματα προς τρίτες χώρες θα πρέπει να γίνει και σε συντονισμό με το, ε, το πού θα βρίσκονται οι καταστάσεις μας. Εσείς αναφέρατε και ε, συστήσατε να αναπτύξουμε ένα τμήμα επιμελητίας με την Αφρική αφενός και με τη Μέση Ανατολή αφετέρου. Θεωρώ ότι ως νομοθέτες θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την πολιτική προς τις τρίτες χώρες που αναφέρεται, κατά 70% να τη στηρίξουμε ε, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Η κίνηση φτάνει στην Ευρώπη από τη Μέση Ανατολή μέσω της Μεσογείου. Θα πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε πολιτικές τις οποίες θα τις προσαρμόσουμε στις ε, ροές της κίνησης. Και όταν θα πρέπει να σκεφτούμε και τις επενδύσεις, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κίνηση προς τις τρίτες χώρες, που σε αυτή την περίπτωση δεν ε, την χάνει της ανάλογης τροφοδότησης και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σύνδεση, διότι εμείς σκεφτόμαστε όλο το σχέδιο αποκλειστικά εντός της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε και εκτός Ευρώπης. Αν δεν παρέμβουμε και εκεί, ελοχεύει ο κίνδυνος να μην υπάρχει διασύνδεση. Ε, αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ε, την πολιτική του τελευταίου χιλιόμετρου, τη σύνδεση δηλαδή του λιμένα με, το, με την ξηρά και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ κύριο Ελκατράου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Ντεολιβέιρα. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η θαλάσσια αυτοκινητόδρομη έχουν ήδη ξεκινήσει και χαίρομαι που κάνουμε έναν απολογισμό. Βλέπουμε τι συνέπειες έχουμε, ώστε να μπορέσουμε να κρίνουμε και τις επενδύσεις μας. Να δούμε αν αυτές οι επενδύσεις ε, οδήγησαν σε αποτελέσματα, αν υπάρχουν συνέπειες για τις ε, ε, ροές των εμπορευμάτων και αν υπάρχουν και συνέπειες στους λιμένες που υποδέχονται αυτά τα εμπορεύματα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε και διάφορα προγράμματα υποδομών αλλά και προγράμματα μηχανοργάνωσης ε, και αντίστοιχα στοιχεία τέτοιου είδους. Θεωρώ ότι όσον αφορά τα προγράμματα υπάρχει υπερεπάρκεια καλών ιδεών. Ε, έχουμε κάποιες ε, άγουσες για κάποια προγράμματα τα οποία είναι αποτελεσματικά και θα μπορούσαμε ίσως να ενσωματώσουμε στο όλο ζήτημα. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως τι συστήνεται για όλες αυτές τις δυνατότητες ε, επενδύσεων. Ποια θεωρείτε ότι είναι προτεραιότητα. Ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να ε, καλύτερα τα κονδύλια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας ή θεωρείτε ότι είναι καλή η κατανομή. Κυρία Μάιστερ για δύο λεπτά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Ολιβέρα για την έκθεσή σας. Σωστό. Είπατε 90, κάποιοι λένε 95% εισαγωγών-εξαγωγών είναι ε, οι ε, εκτός ε, Ευρώπης συναλλαγές και 40% εσωτερικές. Σήμερα δεν έχουμε όρια και σύνορα στα, στη θάλασσα και στις πλωτές μεταφορές, αλλά ένα θέμα είναι η συνεργασία των μεταξύ λιμένων που αναφέρατε. Βρίσκονται σε ανταγωνισμό οι λιμένες και του βορρά εναντί του νότου και μέσα στην ίδια τη ζώνη του βορρά λιμένες βορρά-βορρά ανταγωνίζονται τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τη συνεργασία μεταξύ λιμένων. Κάποια πράγματα λειτουργούν δεν είναι ίσως όλοι ε, ο, ο ένας έναντι του άλλου ανταγωνιστές. Ε, θα μπορούσαν να διασφαλιστούν οι πτυχές της συνεργασίας. Ένα άλλο θέμα είναι και το LNG, ιδιαίτερα όσον αφορά το χώρο της Βαλτικής, ε, διότι ακριβώς όσον αφορά αυτές τις δυνατότητες από το 2015 θα έχουν άλλες οριακές τιμές όσον αφορά το θείο για παράδειγμα. Κατά πόσο βλέπετε εσείς ποια επιρροή μπορεί να ασκήσετε ώστε να διαδραματίζει αυτό ένα ρόλο. Κάποιοι χώροι από πλευρά του ε, δημιουργούν υποδομές για το LNG, για παράδειγμα στην Ολλανδία στα λιμάνια. Είναι μια καλή εναλλακτική λύση για τα λιμάνια του μέλλοντος, μια και είναι πιο καθαρή, ίσως σε αυτή θα μπορούσαμε να εστιαστούμε. Για μια ολοκληρωμένη πολιτική για τις ε, ναυτιλιακές μεταφορές και για τη θάλασσα θα διπλασιαστούν, α το πω έτσι, οι εκπομπέ αυτέ. Αυτό θα διαδραματίζει ένα ρόλο και για την υγεία των θαλασσών κατά πόσον με την κυρία Δαμανάκη αυτό το σας απασχολεί ή, ή δε, μήπως δεν είναι δική σας υπόθεση αυτή. Θα με ενδιαφέρε να το μάθω. Κράμε δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε. Μου λείπει διασύνδεση σε σχέση με την περιοχή του ε, Ρόστοκ είναι μια σημαντική διαδρομή που βλέπω ότι απουσιάζει. Τι γίνεται με το Φέμαν για παράδειγμα εναλλακτικά ε, onshore ε, ε, power supply. Τι γίνεται με αυτή την ενεργειακή κάλυψη. Διότι για παράδειγμα με τις ναυτιλιακές μεταφορές π.χ. και το θέμα της ε, επιβάρυνσης ε, όσον αφορά τις οδικές μεταφορές. Με εκπλήσει ότι δεν υπάρχει διασύνδεση από τη Μεσόγειο ή από την Ελλάδα προς την, ε, τον Εύξηνο Πόντο. ίσως αυτό είναι θέμα που άπτεται και με την Τουρκία π.χ. για παράδειγμα και με τη Βουλγαρία-Ρουμανία, γιατί δεν διαδραματίζει ένα ρόλο ευξήνος πόντος. Ποια προγράμματα, ποια, ε, ποιες πρωτοβουλίες υπάρχουν για ε, short shipping, short sea shipping. Και εδώ, για παράδειγμα, πρέπει να δούμε πώς εσείς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, όχι μόνο η Μεσόγειος και η Βαλτική, αλλά γενικά οι εκπομπές ρήπων να μειωθούν διότι μέχρι σήμερα ε, ε, λειτουργούν χωρίς ε, φίλτρα αυτά τα πλοία στις εγκαταστάσεις τους και ρηπαίνουν το περιβάλλον. Στη Γερμανία έχουμε μια ε, κατάσταση που οι, τα κρατήδια επομίζονται αυτή της πολιτικής. Χρειαζόμαστε όμως ε, ένα ευρωπαϊκό χώρο ε, αρμοδιότητας για τις ναυτιλιακές υποθέσεις και για τα θέματα της θάλασσας. Πώς το βλέπετε αυτό, π.χ. για παράδειγμα στη Γερμανία με την αρμοδιότητα των κρατηδίων δεν υπάρχει εθνική αρμοδιότητα. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ του το συντονιστή κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι θαλάσσιοι αυτοκινητόδρομοι. Ε, είμαι θετικά διακείμενο, αλλά έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω περί τίνο ακριβώς πρόκειται και πού ακριβώς τους εντάσσουμε. Ε, υπάρχουν 40 λιμένες από πλευρά ε, νομοθεσία και προπολογισμού και α, είναι πρόβλημα αυτό. Να σας πω για παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιες πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται για τους λιμένες και τις υποδομές των λιμένων, αλλά οι υποδομές των λιμένων δεν είναι πάντα στραμμένες προς τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους. Από την άλλη έχουμε κάποιες ε, ε, που αφορούν την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, έχουμε κάποιες που αφορούν τη βιομηχανική πολιτική, κάποια στοιχεία που αφορούν ε, την ενεργειακή πολιτική από ό,τι άκουσα και από τον κύριο Καντσιάν μα ενδιαφέρει και το θέμα τη πολιτική γειτονία και τη σχέση με τι τρίτε χώρε και από εκεί και πέρα έχουμε και περιβαλλοντική πολιτική. Και από εκεί και πέρα μα δίνεται και εντύπωση ότι δεν καταφέρουμε να διαβάσουμε με διαρθρωμόνο τρόπο ε, ποια ακριβώ είναι τα προβλήματα. Για να μπορέσουμε να στήσουμε εντό εισαγωγικών αυτόν τον θαλάσσιο αυτοκινητόδρομο θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται και ίσως θα έπρεπε να στραφούμε προς μια διαφορετική ε, κατεύθυνση και να δούμε αν θα είναι πραγματικά ολοκληρωμένο το πρόγραμμα ή αν θα είναι κάτι μεμονωμένο σε κάθε περίπτωση. Και μπορεί να έχουμε έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίος να καλύπτει κάποια στοιχεία ε, πολιτικής ε, θαλάσσιας ε, και κάποια άλλα που να καλύπτει μόνο την πολιτική των λιμώνων και είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα και δεν μπορούμε να βρούμε πού ακριβώς εμπίπτει αυτός ο θαλάσσιος αυτοκινητόδρομος. Η κυρία Γιάλα Σέντερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Ολιβέρα και να τον ευχαριστήσω για την παρουσίασή του. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις ε, επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 τι προοπτικές βλέπετε εσείς ε, βλέποντας τις εργασίες που έχουν γίνει και την πρόοδο αυτών των προγραμμάτων. Εμείς ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση και μας ενδιαφέρει, είναι ανάγκη να εφαρμοστούν και να είναι και αποδοτικά όλα αυτά τα προγράμματα. Υπάρχουν κάποιοι αυτοκινητόδρομοι που θεωρούνται ήδη ότι είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί, ενώ κάποιοι άλλοι χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη. Μπορείτε να μας πείτε εσείς ε, ποιο χρηματοδοτικό μέσο θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση. Κατόπιν, Στι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ, μα ενδιαφέρει να υπάρχουν και συνέργειε με τουλάχιστον δύο ή τρει τομείς, δηλαδή μεταφορέ, ενέργεια και τηλεπικοινωνίε. Θα μπορούσατε να μα πείτε τι γίνεται για παράδειγμα με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, ή την ε, ενέργεια επί της ε, ακτής. Υπάρχουν κάποιες ιδέες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτές τις συνέργειες. Και τέλος, να πω ότι έχω την ίδια αίσθηση με τον κύριο Ρικέ. Είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε σαφέστατα αν πρόκειται για προγράμματα υποδομών, για προγράμματα υπηρεσιών ή για κάτι επιπλέον. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία εγώ από ισπανοϊταλική εμπειρία γνωρίζω ότι έλειπεν ε, σκάφη αρκετά μεγάλου μεγέθους ώστε να γίνεται αυτή η μεταφορά εμπορευμάτων. Μπορείτε να μας πείτε λίγο στο μέλλον πού θεωρούμε ότι εντάσσονται καλύτερα αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ε, <clears throat> πώς βλέπετε κύριε Ολιβέηρα την πιθανή και αν σας έχει απασχολήσει ε, ένας καλύτερος συντονισμός με την Επιτροπή εν ώψη του ότι φαίνεται να ετοιμάζεται μια ε, να υπάρχει μια καινούρια προσπάθεια στα Σκαριά για λιμενική ευρωπαϊκή πολιτική. Και αν είσαστε σε επαφή με την Επιτροπή γι' αυτό, αν βλέπετε ότι υπάρχουν συνέργειες με το θέμα των λεωφόρων της θάλασσας, αυτή είναι μία ερώτηση και η άλλη, εφόσον συζητήσαμε για τοποθέτηση ειδικού συντονιστού για τα ETMS, ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν βλέπατε την ανάγκη να υπάρξει έστω για δύο χρόνια παράταση ή εν πάση περιπτώσει να τοποθετηθεί ένας ειδικό συντονιστής και για τους ε, θαλάσσιους διαδρόμους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ ο κύριος Ντολιβέιρα. Θα θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σε σχέση με τη διασύνδεση με τρίτες χώρες και την επιμελητιακές προσαρμογές σε σχέση με άλλες τρίτες χώρες, πρέπει να πω ότι ασχολήθηκα με αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις επισκέψεις μου στην Ιταλία και στην Ισπανία. Διότι εκείνες οι χώρες, αυτές οι χώρες είναι αυτές που έχουν μεγαλύτερη επαφή με αυτό το θέμα. Ακόμα επισκέφθηκα και μία φορά τον αρμόδιο πρέσβη ε, για την ε, μεσογειακή ε, πτυχία αυτού του προβλήματος και με μεγάλη σπουδαιότητα που δίνεται σε αυτή τη διασύνδεση εξετάσαμε το θέμα. Όμως έχετε δίκιο και κάτι παραπάνω από δίκιο ότι είναι αναγκαίο να μην χάσουμε την ε, δυνατότητα διασύνδεσης που θα μπορούσε να χαθεί αν δεν προαγάγουμε το θέμα και δεν το έχουμε διαρκώς ε, στο επίκεντρο της προσοχής μας. Δεν έχουμε ειδικό μέσο ή εργαλείο γι' αυτό, αλλά τα λιμάνια που εμπλέκονται σε αυτό τη δράση δεν είναι μόνο μεγάλα λιμάνια όπως η Βαλένσια και η Βαρκελόνη, είναι και λιμάνια όπως το Αλικάντε που <clears throat> τίνουν πάρα πολύ σε, αυτή, σε αυτού του είδους τη δραστηριοποίηση και αναφερόμενο σε λιμάνια μπορώ να πω ότι και οι πλειοκτήτες και αυτοί πάρα πολύ ενδιαφέρονται σε αυτή την πτυχή. Δεύτερο, σε σχέση με την τελευταία ας το πω έτσι, δυνατότητα διασύνδεσης ε, εκ του σύνεγγης, last mile. Γι' αυτό δίνω ένα παράδειγμα. Η διασύνδεση στα λιμάνια, στο Όρχους ή στο Γκότεμπεργκ, για παράδειγμα, αποτελούν ε, τμήμα αυτών των ε, υπηρεσιών που στοχεύουν και στα λιμάνια προορισμού και η διασύνδεση μεταξύ ε, επιμελητιακής πλατφόρμας ε, στις δράσεις ε, είναι μέρος των μελημάτων και των ανησυχιών μας. Ακριβώς όταν έρχεται η ώρα να πει κανείς ότι, όταν λέει κανείς ότι αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων που προσπαθήσαμε να καλύψουμε, για παράδειγμα οι επιπτώσεις στο εμπόριο, που είναι ε, και οι επιπτώσεις στο εμπόριο που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας μέσω τόσο πολυσχηδών δράσεων. Είναι αναγκαίο να έχουμε μια γενικότερη επισκόπηση της κατάστασης και τους διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων να τους εντάξουμε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σε σχέση με τέτοιες πρωτοβουλίες. Αλλά πρέπει να πω ότι θα έχουμε και αξιολόγηση επί του τι αλλά πάντα με την λογική που ακολουθήσαμε, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ λιμένος ε, ε εκκίνησης και λιμένος προορισμού όχι μόνο σε σχέση με τις επενδύσεις, τα λιμάνια έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε όλες αυτές τις δράσεις και πτυχές, αλλά και η διασύνδεση με την ενδοχώρα, για παράδειγμα, και αυτή είναι πολύ σημαντική. Και αυτή έτσι αρθρώνεται και τα θέματα ασφάλειας επιπλέον και τα θέματα όρων και προϋποθέσεων στα ίδια τα λιμάνια. Και όταν εσείς φυσικά κυρία αναφέρεστε στη συνεργασία λιμένων, φυσικά αναφέρατε ότι βρίσκονται τα λιμάνια σε ανταγωνισμό. Δεν συνεργάζονται. Μπορείτε να δείτε λοιπόν για την, ε, τα λιμάνια της Βόρειας Αδριατικής και την Ένωση Λιμένων Βόρειας Αδριατικής έχουμε ε, μία προσπάθεια διασύνδεσης, ε, να κάνουμε τα πρώτα βήματα, πράγμα το οποίο είναι ήδη πολύ σπουδαίο. Ε, προσεχώς σε ένα πρόγραμμα Αντριάνος που ε, αναφέρεται στη διασύνδεση από την Ιγουμενίσα της Ελλάδας μέχρι ε, τα λιμάνια της Βόρειας Αδριατικής. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για τη δυνατότητα να φτάνει κανείς στην Ιγουμενίσα και με πληροφορική και τα μέσα της επικοινωνίας να δει κανείς Ποιε ποιες δράσεις ε, ακολουθούνται και τι μπορεί να γίνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κάνοντας αυτό υπάρχει πάντα ο ανταγωνισμός του ενός έναντι του άλλου, αλλά αφρώνονται όλα αυτά μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Βρίσκονται σε ανταγωνισμό διότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία αρθρώνονται εδώ και πρέπει να καταστούν συμβατά και συνεκτικά μεταξύ τους. Μπορεί όμως να επιλεγεί αυτό το οποίο ε, μπορεί να ακολουθηθεί σε σχέση με τις πληροφορίες που αφορούν για παράδειγμα στη διασύνδεση με την ενδοχώρα και τις ε, δυνατότητες ε, διασύνδεσης με την ενδοχώρα, τη διαθεσιμότητα χώρου για τις δράσεις αυτές, στις οποίες, στον οποίο χώρο μπορούμε να καλύψουμε το χώρο αυτό με τις δραστηριότητές μας. Αναφερθήκατε επίσης στο LNG. Το LNG ήταν μια έκπληξη, διότι ξέρετε σε σχέση με την Βαλτική και την Βόρεια Θάλασσα μέχρι το 2015 θα πρέπει να υπάρξουν οι δράσεις ώστε να ε, συμμορφωθούν όλοι με τους κανόνες ΣΕΚΑ. Δηλαδή 0,1% περιεκτικότητα θείου για, αυτά τα, ε, για τα καύσιμα και τις εκπομπές. Ε, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό να μετατεθεί αυτό και να μπορέσει να λειτουργήσει και για άλλου είδους καύσιμα. Ήδη έχουμε την πρόθεση να αντιμετωπίσουμε ένα εγχείρημα, ένα πρόγραμμα με μεθανόλη και το LNG φαίνεται ότι θα είναι το πιο σημαντικό καύσιμο για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και δράσεις. Ήδη στη Βαλτική έχουμε ένα πρόγραμμα που αφορά την διασύνδεση και των ε, ε, λιμένων ανεφοδιασμού, bunkering. Απόλυτα κατανοητό αυτό διότι ανησυχούν για την κατάσταση στη Βαλτική, επειδή η Βαλτική όπως γνωρίζετε είναι μια κλειστή θάλασσα, δεν ανανεώνεται και δεν οξυγονώνεται και αυτό, αυτές οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν. Και άλλα καλά μαντάτα είναι ότι υπάρχει η πρόθεση να αναπτυχθούν νέες διευκολύνσεις και μέσα σε, ε, ε με τον συνδυασμό την, την διασύνδεση ε, Ρότερνταμ και Γκότεμπορκ. Και αυτό είναι πολύ καλά ε, μαντάτα για το τι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τομέα. Έχετε όμως δίκιο και υπογραμμίσατε το θέμα της ε, υγείας στη θάλασσα. Σίγουρα το θέμα αυτό είναι, έχει κομβική σημασία. Είναι μία από τις επιπτώσεις όσον αφορά την χρήση πιο καθαρών καυσίμων. Άμεσα ε, έχει επιρροή στην υγεία και την ποιότητα σε σχέση με τη θάλασσα. Αναφερθήκατε κύριε Κράμερ για το Ρόστοκ και τη διασύνδεση και σε σχέση με την Κτίνια ε, που ε, ξεκινά ας το πω έτσι ε, στις 28 Νοεμβρίου, ε, μεθαύριο δηλαδή, σε δύο μέρες. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η στοχοθέτηση και αυτή η πρόθεση να προχωρήσει αυτό. Είναι ένα από διάφορα προγράμματα ε, πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών που στη συγκεκριμένη φύση αυτών των δράσεων αναφέρθηκα στην αρχή. Φυσικά έχετε δίκιο. Ενδιαφέρον θα ήταν να είχαμε ένα ευρύτερο ε, ένα ευρύτερο φάσμα διασυνδέσεων μεταξύ π.χ. Ε, του εύξηνου πόντου και της Μεσογείου. Όμως πρέπει εδώ να σας πω ότι προσπάθησα κατά την ε, επίσκεψή μου στον πύργο Μπουργκάς της Βουλγαρίας προσπάθησα να διατυπώσω αυτό το ζήτημα, το ερώτημα σε σχέση και με την διασύνδεση Μπουργκάς πύργου Αλεξανδρούπολης διότι κατανοώ πάρα πολύ καλά ότι ο Βόσπορος είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή είναι τα στενά πάρα πολύ ευαίσθητα και πρέπει να κατανοήσουμε την ανησυχία που έχουν οι Τούρκοι όσον αφορά την αύξηση του όγκου μεταφορών με τα δεξαμενόπλια που διασχίζουν τον Βόσφορο από τα Δαρδανέλια, από το Αιγαίο προς τη Μαύρη Θάλασσα και τούμπαλιν από τη Μαύρη Θάλασσα προς το Αιγαίο, προς τη Μεσόγειο. Υπάρχει εδώ διασύνδεση, διότι η διασύνδεση προφανώς μεταξύ πύργου Μπουργάς και Αλεξανδρούπολης ε, αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες επειδή διασχίζει περιοχή προστατευόμενη από το δίκτυο Natura 2000. Όμως, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτή τη διασύνδεση, αυτόν τον άξονα, διότι καλό θα είναι και για τη Βουλγαρία αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης ευρύτερα. Σε παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο, ναι, λέει ο μιλητής, ναι. Αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις δράσεις σε ένα ε, ενιαίο ολοκληρωμένο πλαίσιο να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια ολοκλήρωσης. Θα συνεχιστεί σίγουρα. Αναφέρθηκα πιο πριν και είπα ότι προσπαθούμε προς την κυρία Αγιάλα αυτό και το είπα πιο πριν. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τους κύριους ε, άξονες τις τα κυριότερα χρηματοδοτικά, χρηματοοικονομικά μέσα για αυτές τις δράσεις. Καλύτερο πιστεύω θα ήταν αν θα μπορούσαμε να ε, επιλέξουμε τα, τις επιμέρους συνιστώσεις για την χρηματοοικονομική κάλυψη από πλευράς των ετούντων για παράδειγμα. Αλλά έχετε δίκιο. Είναι ανάγκη να ταυτοποιήσουμε και να εντοπίσουμε αυτού του είδους ε, τα ε, οχήματα, τα πλοία, τα οποία θα πρέπει να είναι τα πιο ενδεδειγμένα για τις ανάγκες μας και όχι να δημιουργούν ε, προβλήματα. Τελευταία ερώτηση είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό σε σχέση με τις ε, διάφορες ε, λιμενικές πτυχές, ξεκινώντας από τους ε, ορισμούς για παράδειγμα για αυτούς τους λιμένες, προσπαθώντας πάντα να δημιουργήσουμε παρόμοιες διασυνδέσεις με κοινού είδους ε, επαφές και ε, διασυνδέσεις και επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών λιμένων. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, πράγματι είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στη Βαλτική. Παρακαλώ, έχετε και εσείς 10 λεπτά κύριε Τελίνκα. Πρώτα ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Σας διαβεβαιώθαμε σήμερα γιατί έχω αρχίσει σήμερα να βραχνιάζω και δεν θα αντέξω να μιλάω για 10 λεπτά. Ξεκινώ πάντως με μία σύντομη επισκόπηση των συνθήκων που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να πέρασω πιο συγκεκριμένα σχόλια. Τους τελευταίους 12 μήνες ε, σημειώθηκαν ε, εξελίξεις, πρόοδο σταθερή, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Προχωρήσαμε σταθερά προς τα μπρος, με όλα τα θετικά και τα αρνητικά. Και για πρώτη φορά πρέπει να σημειώσουμε ότι είχαμε αναγνώριση της ε, οικονομικής ανάπτυξης που θα φέρει η Βαλτική που αφορά όχι μόνο τη Βαλτική και την Πολωνία, αλλά από, από τους, ε, πολλές από τις χειροπεριοχές, κεντρική Ευρώπη. Φερρυπίν, η αυτοκινητοβιομηχανία της κεντρικής Ευρώπης θα ήθελε περισσότερη, ε, περισσότερα ποσοστά στις μεταφορές της υδροδρομικές, από 50% σε 60%. Για δε την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την πατρίδα μου και τη γειτονική μας χώρα, τη γείτονα χώρα που είναι και μεγαλύτερη παραγωγός αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Ε, παραδείγματα έχουν τέτοια αιτήματα. Η Φιλανδία, από την άλλη που έχει παραγωγή ξυλίας και χαρτοπολτού ενδιαφέρεται επίσης για τις ε, ε, θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων για τα προϊόντα της. Αυτές είναι οι θετικές εξελίξεις. Επίσης ως προς θετικές εξελίξεις μπορώ να αναφέρω σημαντική σημαντικό ενδιαφέρον και στράτευση από τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. Επί παραδείγματι, η Πολωνία δραστηριοποιείται ιδιαίτερα και εντατικά. Ωστόσο, Ακόμη παραμένουν τα προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν, τα εθνικά συμφέροντα που τείνουν να υπερέχουν των κοινών ευρωπαϊκών συμφερόντων, του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος, κατά κανόνα, αλλά βλέπουμε και κάποιες ε, αρχές οι οποίες είναι διατεθειμένες ε, να προβάλλουν το ευρωπαϊκό συμφέρον, κυρίως στις σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης της Ευρώπης. Βλέπουμε επίσης τα βραχυπρόθεσμο συμφέρον να επικρατεί στα θέματα της ε, διασυνδεσιμότητα στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης ή μάλλον έχουμε την αίσθηση ότι ορισμένες φωνές πολιτικές ε, διεκδικούν ε, την πατρότητα του χρήματος που διατίθεται και άρα και τον προσδιορισμό της χρήσης του. Βέβαια, στην Ευρώπη τη σύγχρονη εποχή που έχουμε πει, αυτά είναι όλα αυτονόητα. Αλλά παραμένουν και τα προβλήματα του παρελθόντος παρά την γενική σταθερή και καλή πρόοδο που σημειώνεται. Συγκεκριμένα τώρα, και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ ξεχωριστά σε δύο θέματα. Όταν ξεκινήσαμε πριν από δέκα περίπου χρόνια, ε, προσπαθούσαμε, ε, μάλλον είχαμε την τάση να ακούμε από τους πολιτικούς ε, ότι θα υπάρχει ταχείας, ε, μεγάλης ταχύτητας ε, τρένο από το Ταλίν ε, μέχρι την Βαρσοβία. Τώρα προσπαθούμε να του εξηγήσουμε ότι τα όνειρα αυτά δεν υλοποιούνται από την μια μέρα στην άλλη και χρειάζονται υποδομές. Έχουμε φτάσει ωστόσο στην εποχή που πρέπει πια να επικαιροποιήσουμε την γραμμή που έχουμε στη διάθεσή μας ήδη και εδώ θα σας πω ποιες είναι οι δυσκολίες. Και δεύτερον, δεύτερη διάσταση, μέλλον, το λεγόμενο Baltica 2, εγώ έτσι θα το ονόμαζα, και μια νέα γραμμή που θα συνέδεται το Ταλίν με τη Βαρσοβία. Υπό την επιφύλαξη βεβαίω τη έγκριξη από τα ευρωπαϊκά ε, όργανα, θεσμικά όργανα που ήδη έχει εγγραφεί στη γραμμή Βαλτική-Αδριατική. Αυτό που, διαβλέπουμε λοιπόν είναι υποστήριξη από τους Πρωθυπουργούς και Υπουργό των Μεταφορών που δόθηκε πέρυσι στο νέο αυτό σχέδιο έχουμε νέο επίπεδο επικοινωνίας και εργασίας με μια task force που θεσπίστηκε και συγκεκριμένα συναντήσεις των υπουργών των μεταφορών με κατά πάσα πιθανότητα μια, τον Ιανουάριο μια μελέτη που αναμένεται ώστε να δούμε τι θα πρέπει να καλύπτει αυτός ο νέος φορέας που θα εποπτεύει το όλο σχέδιο. Αυτό νομίζω θα είναι η απο... Το, το, το κρίσιμο σημείο. Η Εστονία που θα ορίσει πιστεύουμε και τον μειοδοτούντα σε μερικές εβδομάδες όπως και η Λιθουανία και η Λετωνία που θα ακολουθήσουν αργότερα, ήδη δίνουν καλές κατευθύνσεις. Η Πολωνία, όπως είπα, ε, διαδραματίζει ενεργό ρόλο. Μέχρι τώρα αυτή είναι η κύρια δέσμευση που σημειώνουμε. Και οι Φιλανδοί βέβαια που επανακάμπτουν. Είναι πολύ ενθαρρυντική η στάση τους. Πάντως, τώρα έχουμε μια νέα προσέγγιση, 35 χιλιοστά γραμμή. Αλλά ποια είναι η κατάσταση με την ε, τωρινή κατάσταση και με την ισχύουσα γραμμή για να δούμε την κατάσταση. Η Εστονία παρουσιάζει μια καθαρή εικόνα. Δεν ήταν εύκολο να συμφωνήσουμε στα κύρια θέματα από την αρχή με την Εστονία, όμως τώρα έχει προχωρήσει σημαντικά ε, και ως εκ τούτου η Εστονία δεν ε, να δυσκολεί. Η Λετωνία, που ίσως να θυμάστε λόγω της οικονομικής κρίσης χρειάστηκε να αναβληθεί για 1,5 περίπου χρόνο τις εργασίες, αλλά ξανάρχισαν τώρα και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά σε επίπεδο Ρήγα. Για την ε, Λετωνία θα θυμάστε ότι η ενσωμάτωση της Ρήγα ήταν πάρα πολύ σημαντικός παράγων ε, και χάρη σε αυτό τώρα έχουμε την υποστήριξη των Λετωνών. Η Λιθουανία έχει ακόμα εκρεμεί ζητήματα προγραμματισμού που μας έχουν καθυστερήσει σημαντικά ως προς την διπλή τροχιά. Θα θυμάστε ότι είχαμε χρησιμοποιήσει την αρχική τροχιά, την ρωσική, και το, τη χάραξη που έχουμε για να φτιάξουμε μια παράλληλη διπλή τροχιά, παράλληλη με τη ρωσική. Αυτά τα προβλήματα τώρα σχετίζονται προφανώς και με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση μετά τις εκλογές θα χρειαστεί να δώσουμε νέα όθηση στα προβλήματα, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Και με τη Λιθουανία, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα σημειωθούν καθυστερήσει. Η Πολωνία. Η Πολωνία έχει μία λεπτή, ε, μία λεπτομερή κατανομή για την ε, παρέκκληση από τον ΕΛΚ που είχε προβληθεί όπως θα θυμάστε. Θα κοιτάξουμε να σωματωθεί στις ε, δημοσιονομικές προοπτικές αλλά πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθεί και έχουμε και μελέτες σχεδιασμού που φτώνει μέχρι το Σουάλκι. Πρώτα δεν θα επαναλάβω τόσο έχουμε περιλάβει στην εκθεσή μα. Τα κύρια σημεία μόνο θέλω να υπογραμμίσω. Ότι δηλαδή τηρούμε το χρονοδιάγραμμα, Λίγες καθυστερήσει έχουμε, κάποιε δυσκολίε σημειώνονται, αλλά πάντω μπορούμε πιστεύουμε μέχρι το τέλος και ενώπιση των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών να είμαστε έτοιμοι και γίνεται πολλή δουλειά για, την, για το νέο σχεδιασμό 1435. Για την Βαλτική μπορούμε να πούμε ότι η αντίληψη που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις κατευθυντήριες γραμμές και το Connecting, Europe Connecting ε, ως μέσον, ε, νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική. Θα μπορούσα να σας δώσω πολύ λεπτομερή στοιχεία με τον αριθμό των στενοπών που σημειώνονται. Το μόνο μπορώ να πω είναι ότι από την Επιτροπή των Μεταφορών είχαμε πάντοτε υποστήριξη, από, από εσάς δηλαδή είχαμε πάντα υποστήριξη για το πακέτο αυτό, για τις προσπάθειες αυτές. Πρόκειται για μια πτυχή που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε βεβαίως με θάρρος, αλλά στη τελευταία ανάλυση αποτελεί μια από τις προκλήσεις του, της εποχής. Για τα 10 δις από το Ταμείο Συνοχής δεν θέλω να πω δύο λόγια γιατί πρέπει να σωματωθούν, για, το θέμα του αν θα πρέπει να σωματωθούν στο Europe Connecting. Περιμένω τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουμουτσάκος δύο λεπτά γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και σας παρακαλώ να είστε σύντομος κατά το δυνατόν. Πίσω τα δύο λεπτά. Ε, εγώ διαπιστώνω με χαρά και ικανοποίηση ότι η εκτίμηση είναι ότι τα πράγματα ότι τα πράγματα ε, αναπτύσσονται με τρόπο ικανοποιητικό. Το επανέλαβε ε, ο συντονιστής πολλές φορές στην εισήγησή του. Αλλά βεβαίως αυτή η θετική εικόνα δεν είναι 100% πιστική γιατί θέλαμε να ακούσουμε και ποια είναι τα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζετε τώρα. Ποια είναι τα βασικά σας προβλήματα. Αν μπορούσατε να ιεραρχήσετε δύο ή τρία για να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Είναι πολύ θετικό ότι έχουμε μια θετική πρόοδο, αλλά θα ήθελα πραγματικά να ακούσω αν μπορούσατε να κάνετε μια ιεράρχηση των δύο-τριών προβλημάτων που σας απασχολούν περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λιμπεράτσχη για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά άκουσα την παρουσίασή σας σήμερα. Έχω βέβαια κάποιες ερωτήσεις. Ε, καταρχάς, το 2013 που θα ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο. Τι ακριβώς εννοείται με το πρώτο στάδιο. Δεύτερον, αναφερθήκατε στην Ιστονία, τη Λιθουανία και τη Λετωνία, οι οποίες έχουν μια κοινοπραξία και λέτε ότι θα ήταν λογικό να επεκταθεί και στην Πολωνία. Ισχύει αυτό. Τρίτον, λέτε ότι το πρώτο στάδιο προϋποθέτηση και την ε, ε σιδηροδρομική γραμμή μέχρι το Πιελοστόκ και τη γραμμή Βαρσοβία-Πιελοστόκ. Λέτε επίσης ότι παίρνουμε κονδύλια από το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2012, αλλά εγώ από ό,τι βλέπω Έχετε μία γραμμή 14-35 χιλιοστά και από πού θα προέρχεται η χρηματοδότηση όμως για τη Λετωνία και τη Λιθουανία ε, όλη η σιδηροδρομική γραμμή προσαρμόζεται σε αυτό το άνοιγμα τροχών. Επίσης, τι γίνεται με την πρόοδο στην Πολωνία και όταν θα προσθέσουμε και το βασικό δίκτυο της Βαλτικής, τι χρηματοδότηση θα δοθεί σε αυτό. Αν ε, κατάλαβα καλά, το πιο εύκολο θα ήταν να έχουμε κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής. Ευχαριστώ, κύριος Κράμερ, για δύο λεπτά. Um, καλά, κυρία Μάισνερ πρώτα, παρακαλώ, δύο λεπτά. Ναι, ναι, ε, κοιτάξτε. Είναι ένα καθοριστική σημασία σχέδιο, γιατί Μπορεί ο καθένα να λέει ότι είναι ωραίο ότι μπορούμε να μπορούμε να ταξιδεύουμε με τον σιδηρόδρομο να την Ευρώπη, αλλά από τη Βαλτική στην, υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει σύνδεση. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν το use it or lose it, αυτή η αρχή βλέπετε να ε, θέτει σε κίνδυνο το σχέδιο Baltica. Βλέπετε κάποιο κίνδυνο μέσω αυτού. Το The Mason Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη. Ε, θα μπορέσει να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τη διασύνδεση με την Πολωνία που αναφέρατε. Και τώρα που περικόπτονται τα κονδύλια βλέπετε κίνδυνο για την υλοποίηση του έργου. Νομίζω ότι είναι σαφής η ερώτηση μου. Και η απάντηση νομίζω ότι είναι σαφής, αλλά έπρεπε να τη διατυπώσω. Καλώ, ο κύριο Κράμαρ τώρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχά, ευχαριστώ πολύ για το, για το έργο σα, για τι προσπάθειέ σα. Η Λετωνία και η Λιθουανία θα είναι έτοιμε στο 2014. Το, η Πολωνία για το Σοβάλκι με Χρυτομπίλστοκ ε, είναι η προβληματική διασύνδεση. Για το 2020 προβλέπεται. Ναι, ναι, έτοιμη. Ε, μα είπατε νωρίτερα, μα είπε μάλλον νωρίτερα η κυρία Πάη ότι δεν έχουμε πρόβλημα τα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν, αλλά από την άλλη Υπάρχει σε αυτό το θέμα δυσκολία στι διασυνδέσει αυτέ στην Πολωνία και γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2020 μέχρι να κλείσει αυτό το κενό στη διασύνδεση στη δεδρομική αν όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι νωρίτερα, γιατί πρέπει να καθυστερήσουν αυτά τα έργα. Και γιατί πρέπει να περιμένουμε από το 2014 μέχρι το 26 χρόνια για να φτάσουμε μέχρι την ε, Πολωνία και οι μεταφορές, μιλάτε για μεταφορές εμπορευμάτων φαντάζομαι, αλλά των επιβατών. Οι επιβατικές ε, μεταφορές είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικέ. και εγώ που ταξίδεψα μια φορά από το Βερολίνο μέχρι το Ταλίν της Εστονία με το τρένο, Έκανα 60 ώρες το δρόμο, 60 ώρες το τρένο. Φαντάζομαι ότι ένας επιβάτη δεν θα αντέξει να κάνει αυτή τη διαδρομή. Άρα όταν θέλουμε να κάνουμε και επιβατικές μεταφορέ, πρέπει να είναι πολύ πιο σύντομα και άνετα τα τρένα. Αχ, τι ωραία πράγματα μας λέτε, λέει ο κύριος Σίμψον, ο κύριος Ρόμπερτ Τζέλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. šī projekta ietveros. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα τεχνικό, θα το λύσουμε αμέσω. Θα τα πω στα αγγλικά, ναι, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχάς τον συντονιστή για τα σχόλιά του. Δύο ερωτήσεις. Τι σκέφτεστε για την κατάσταση για κάποια από τα κράτη που συμμετέχουν στο Βαλτική 2. Ε, κάποιες ε, χώρες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή θα συμμετέχουν. Ε, θα υπάρχει ίσως σύνδεση Ρήγα μέχρι τη Ρωσία ή θα υπάρξει και κάτι ε, πολιτικής γειτονίας για να υπάρχουν επενδύσεις σε ρωσική επικράτεια. Και από εκεί και πέρα δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα για τις, ε, ε, τα επόμενα 7 χρόνια, τις επόμενες δημοσιονομικές προπτικές. Ε, θεωρείτε ότι είναι πιο ε, μικρότερες, πιθανότητες, μικρότερες πιθανότητες να έχουμε επενδύσει εκεί. Υπάρχει και μια μελέτη σκοπιμότητας ε, για ε, ηλεκτροκίνηση στην ε, κατεύθυνση Ανατολή προς Δύση και γι' αυτό θα χρειαζόμαστε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα σχολιά σας λοιπόν επ' αυτού. Επίσης, θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να μελετήσουμε το μέλλον της Βαλτικής ως ένα ε, πρόγραμμα διπλής τροχιάς. Υπάρχει δυνατότητα να εξετάσουμε κάτι τέτοιο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ε, τις ε, δυνατότητες που έχουμε εδώ για το 15-20 άνοιγμα και 14-35. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο να απαντήσετε κύριε Τέλικα. Αν μπορέσετε και σε 10 λεπτά θα με βοηθήσετε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω τι μπορώ. Θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω. για την ταξινόμηση των προβλημάτων. Θα είναι ένα μείγμα. Αφενός έχουμε το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε μια περιοχή όπου, όπως και σε κάποια άλλη μέρη της Ευρώπης, δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, δηλαδή δεν υπάρχει σταθερότητα στην κυβέρνηση όπως θα θέλαμε. Με κάθε αλλαγή κυβέρνησης, κάθε φορά έχουμε καθυστερήσει με τις κυβερνήσεις συνασπισμού πάντα έχουμε νέα στοιχεία που εισάγονται στα προβλήματα. Αυτό όμως είναι πολιτική, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά από αυτού. Είναι όμως κάτι το οποίο περιπλέκει τη ζωή μας αρκετά. Όσον αφορά τώρα τα πιο πρακτικά προβλήματα. Ακόμα προσπαθούμε να μειώσουμε ένα δυσανάλογο ε, στοιχείο που είχαμε, ε, το γεγονός ότι θέλαμε να έχουμε στην αρχή στη Βαλτική όλα τα, ε, όλες τις χώρες και απ' την άλλη σε κάποιες από αυτές τις χώρες θέλαμε να εξετάζεται ο σιδηρόδρομος της Βαλτικής ως ένα τμήμα περαιτού ανταγωνισμού. Το έχω πει και στο παρελθόν και θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό, σε κάποιες ιδεοδρομικές επιχειρήσεις ε, δραστηριοποιούνται εντός ε, της χώρας τους ως μονοπόλια. Και για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι συγκεκριμένε συμπεριφορέ τι οποίε πρέπει να εξετάσουμε. Το θέμα οργάνωση σε πρακτικού όρου λοιπόν εξακολουθεί να δημιουργεί πρόβλημα. Επίση υπάρχουν θέματα άλλα, όπω για παράδειγμα η καθυστέρηση στο σχεδιασμό. Υπάρχουν επίσης ε, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κάποιες άλλες μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν ότι γίνονται μελέτες για χι εκατομμύρια ευρώ, μετά έχουμε ύφεση και πρέπει να δούμε άλλες εναλλακτικές λύσεις και εξετάζουμε το θέμα της διπλής γραμμής. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να εντοπίσουμε κάποια προβλήματα. Πάντα είναι ένα συνδυασμό προβλημάτων και από χώρα σε χώρα αλλάζουν. Τώρα, Γι' αυτό το λεγόμενο πρώτο στάδιο, σας παρακαλώ μην τα παίρνετε κατά γράμμα αυτά που σας λέω. Ε, το 1435 άνοιγμα είναι κάτι το οποίο πάντα το είχαμε κατά νου. Ε, κάνουμε αναβάθμιση μέχρι το 15-20, η οποία λίγο πολύ θα γίνει μέχρι το τέλος αυτών των δημοσιονομικών προοπτικών υπάρχουν και κάποιες στενοποί τις οποίες γνωρίζαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε, όπως για παράδειγμα την απόφαση της Πολωνίας για το κατά πόσον θα υπάρξει παράκαμψη ή όχι. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το επιλύσουμε και το γνωρίζαμε, το ξέραμε ότι θα περάσει στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Το είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν. Και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι πολωνικές αρχές θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπίσει το θέμα με διαφορετικό χρονικό ορίζοντα. Ε, πλέον όμως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αρκετά γρήγορα. Υπήρξε μια ερώτηση για την Πολωνία και τις ε, χώρες της Βαλτικής, αν μπορεί να, να εντάξουμε και την Πολωνία εδώ. Ο, ε, όπως σας είπα, η Πολωνία συμμετέχει ενεργά, συμμετέχει και στην Task Force. Προς το παρόν βέβαια δεν μπορώ να περιμένω πολλά περισσότερα από την Πολωνία από όσα κάνει αυτή τη στιγμή. Επομένως, ναι, ε, το Rail Baltica 2 αφορά και την ε, Πολωνία, αλλά υπάρχει και μια νέα γραμμή στη Βαλτική. Ε, στην Πολωνία δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει αλλαγή στο διάδρομο, αλλά ποτέ δεν ξέρετε και τι μπορεί να συμβεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση, η Πολωνία αποφάσισε να χρηματοδότησει την ε, ε, αναβάθμιση από το Ταμείο Συνοχής. Ε, δόθηκαν τα κονδύλια. Η επαρκής χρηματοδότηση βέβαια σημαίνει ότι η Πολωνία αποφάσισε να κάνει περισσότερα πράγματα με το ίδιο ποσό χρημάτων. Μπορεί να μην περάσει σε γραμμές υψηλής ταχύτητας, αλλά θα αναβαθμίσουν στο ε, σε άλλο άνοιγμα τροχών και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει και τη στάση... Σε σχέση με τη στάση των Πολωνών, η πρόοδος στην Πολωνία νομίζω είναι σαφές. Σε σχέση με τη γραμμή αυτή και την ε, ε, ανάπτυξη της έχει, υπάρχει μια μελέτη από πρεβάς Σουβάλκη και τώρα έχουμε μια καλή, ας το πω έτσι, ανάλυση των επιμέρους δράσεων που πρέπει να γίνουν για και την χρηματοδότηση και την παράκαμψη και αν όλα αυτά υλοποιηθούν για την ε, βαλτική αυτή διαδρομή τότε πιστεύω ότι θα έχουμε δυνατότητα να προχωρήσουμε και να δούμε και τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Υπήρξε μια ερώτηση για τη χρηματοδότηση, για τη νέα γραμμή. Αυτό πρέπει να το δούμε ακόμα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση της μελέτης των μελετών. Μπορεί να έχουμε από το 2,5-2,8 ή και τα 4 δις ευρώ. Εξαρτώνται αυτά τα ποσά από ε, πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Και υπήρξε μια ερώτηση αν θα μπορούσε να υπάρξει μια γενικότερη εναλλακτική ε, διαδρομή θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα ε, μέρη αυτά και αυτό είναι εκείνο το οποίο θα μας κάνει να περάσουμε από το 2,5 ίσως το 2,8 ίσως και μέχρι τα 5 δις ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν μετά τα, ε, από πλευράς των ε, θεσμικών οργάνων να υπάρξει συγχρηματοδότηση. Είναι σημαντικό όταν κάνουμε λόγο για μια οικονομία που αντιμετώπισε στο παρελθόν πολύ δύσκολες περιόδους ε, κάνοντας λόγο για ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό εγχείρημα ε, ευρωπαϊκής ε, σημασίας και σε σχέση και με την περιοχή της Βαλτικής κάνουμε λόγο για περιορισμένο αριθμό ε, κατοίκων σε σχέση με τις ε, επιβατικές μεταφορές ε, παρότι έχει σπουδαίο ρόλο η πτυχή αυτή. Αφήνουμε στο περιθώριο το θέμα της μεταφοράς επιβατών αλλά σε σχέση και με τη Ρήγα έχει την σημασία του για προτάσεις που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για την Δυτή διαδρομή από το Καλίν στη Βαρσοβία, μια διαδρομή, θα ε, λειτουργούσε με απώλεια και θα έπρεπε να ε, επιδοτείτε, να επιχορηγείτε. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι μπορεί να, ήταν, ε, να υπήρχαν διαφορετικές καταστάσεις στο παρελθόν. Θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να πορευθούμε με σύμνοια για να μπορέσουμε να ε, δημιουργήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Για τις τελευταίες ε, ερωτήσεις ε, που διατυπώθηκαν δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα απόλυτα την ερώτηση σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα υπό τον όρο της έγκρισης που θα προαπαιτεί το Ήδη κάνουμε λόγο για ένα νέο εγχείρημα σε σχέση με τη Βία Μπάλτικα και δίνεται μια νέα διάσταση σε αυτό. Τώρα υπήρξε και μια άλλη ερώτηση σε σχέση με το αν θα διακυβευτούν αυτά τα προγράμματα. Δεν νομίζω. Φυσικά βλέποντας τη σημερινή, τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων είναι πολύ νωρίς να πει κανείς και να προδικάσει τι θα γίνει και με την ε, ε, νέα αυτή πορεία, τη νέα γραμμή και ποιες δράσεις θα πρέπει να αναλυθούν για σημαντικές ε, αλλαγές της ε, ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλαγή του συνολικού προγράμματος, τότε θα μιλούσαμε πράγματι για διαφορετική προσαρμογή και θα μιλούσαμε και για διαφορετική κλίμακα χρηματοδότησης για μια νέα τέτοια γραμμή. Αυτό είναι σίγουρο θα μπορούσα να πω, αλλά αυτό είναι κάτι επί του οποίου δεν θα ήθελα να κάνω κάποιες εικασίες. Και τέλος, στην ερώτηση Ζήλα. Εγώ πάντα Προσπαθώ να είμαι έντιμος και ακέραιος σε σχέση με τις συζητήσεις με τους υπουργούς των βαλτικών χωρών, λέγοντας ότι η Βία Μπάλτικα είναι πράγματι ευρωπαϊκή προτεραιότητα λόγω της ε, εμβέλειας αυτού του εγχειρήματος. Πρέπει να υπάρξει συνέργεια μεταξύ του άξονα βορρά-νότου, ανατολής-δύσης, σίγουρα. Αλλά δεν θα έπρεπε κανείς να αναμένει κάτι το πιο ξεχωριστό, για παράδειγμα σε σχέση με τον άξονα Κάουνας Ρίγα. Θα πρέπει να βασιστούμε στην δημιουργία συνέργειας που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Το άλλο σε σχέση με τη Ρίγα είναι η ένταξη της ε, Ρίγας μέσα στις ε, διασυνδέσεις αυτές υπό την ε, πτυχή της συνιστώσας Ανατολής Δύσης, διασύνδεσης μεταξύ του άξονα Ανατολής Δύσης. Έτσι θα ήθελα να απαντήσω στο, στην παρέμβασή σας. Και για την τελευταία ερώτηση, αν βλέπω να διακινδυνεύει η βία Μπάλτικα με την χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων ή πρωτοβουλίων. Όχι, δεν θα διακινδυνεύσει αν είμαστε συνετοί και προσαρμοστούμε σε αυτά τα οποία απαιτεί η ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτή την κλίμακα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι με την έγκριση αυτού του πακέτου της δέσμης μέτρων ευελπιστώ ότι θα μπορέσει να προχωρήσει η Βία Μπάλτικα και να αναβαθμιστούν οι ε, κορμοί διασύνδεσης με την Βία Μπάλτικα υπό τους όρους ε, ε, των μεταφορών και για το θέμα της επιμελητιακής ε, συνδρομής και υποστήριξης απευθύνω έκκληση στους ευρωβουλευτές για τη Βία Μπάλτικα να αντιληφθούν ότι αυτά τα λογιστικά κέντρα θα πρέπει να ενταχθούν μέσα σε ένα ολοκληρωμένο τέτοιο πρόγραμμα και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό και από πλευρά χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βαλέντιντο Ολιβέρα, κύριε Βίνκ, ε, κύριε Τελίκα για τις απαντήσεις σας. Εδώ σε ευχαριστώ και την κυρία Πέις που χρειάστηκε να αποχωρήσει. Ξέρετε ότι μια φορά το χρόνο κάνουμε τις συναντήσεις, αύριο θα ακούσουμε και τους λοιπούς συναδέλφους σας. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες ε, οι παρατηρήσεις σας για τους συναδέλφους της Επιτροπής. Και βεβαίω όποιο θέλει μπορεί να πάρει το, ε, ένα αντίτυπο τη εκθέσεω, το βλέπετε εδώ δίπλα. Okay, colleagues, the next item that we need to... Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τώρα να δούμε το θέμα των του ελέγχου των ε, λιμένων, εκτός ελέγχος λιμένων, έλεγχος των λιμένων από το κράτος, των πλοίων από το κράτος λιμένα. Δική μου τροπολογία, 24 τροπολογίες πέραν των όσων έχω εγώ καταθέσει. Συνεδρία των συντονιστών πρέπει να γίνει στις 14 Νοεμβρίου. Έγινε στις 14 Νοεμβρίου για να συζητήσουμε τα θέματα και να δώσουμε κίνητρα στα κράτη τη σημαία να, να κυρώσουν τις σχετικές διεθνεί συμβάσεις. Ωστόσο, ειδικότερα για τα μικρότερα κράτη-μέλη, και ανησυχία ότι ίσως υπερβολικέ νίωψει ε, να είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Ύστερα από τις διαπραγματεύσεις λοιπόν με το Συμβούλιο ιδιαίτερος προτείνω να καταλήξουμε επί της αρχής τώρα για το πεδίο των ε, αποφάσεων που θα προκύψουν ύστερα από περαιτέρω διαπραγματεύσεις με μια ρήτρα σοφή ότι δεν θα πρέπει να ε, αναλυθεί η παραμικρή πρωτοβουλία μέσω της νέας ε, σύμβασης για τους εργάτες θάλασσας ώστε να υπονομευθεί η ισχύους ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφερόμαστε ειδικά στις συμβάσεις περί εργασίας θάλασσα, αλλά και λοιπές συμβάσεις που αφορούν τις νεοψίες. Η ΔΕ Επιτροπή των Μεταφορών ξέρουμε ότι πάντοτε πίεζε για πιο αυστηρές διατάξεις, όχι για υποβασμό του παιδού. Και στόχος μας είναι να μην στοχεύσουμε συγκεκριμένα κράτη-μέλη που ενδεχομένω έχουν καθυστερήσει την κύρωση, αλλά εκείνα τα κράτη-μέλη όπου γνωρίζουμε ότι είναι παράδεκτε οι προποθέσει και προδιαγραφέ και μπορεί να προξενούν κινδύνου ασφάλειας. Όταν λοιπόν είναι κακό το επίπεδο των νιουψιών από το κράτο του λιμένα, θα πρέπει ιδιαίτερω να εντοπίζονται τα καράβια αυτά. Το ΕΛΚ ξέρω ότι ως προς την τοποθέτηση αυτή διαφοροποιείται. Αλλά όπως είπα, είναι απαραίτητο πιστεύω να είναι η θέση μας ισχυρή και ενωμένη στις διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Επίσης, εγγύησεις για την εφαρμογή της, ε, με, της τροποποιημένης οδηγίας προς τις, ε, τους ελέγχους ε, του κράτους λιμένα με τις νέες συνθήκες που θα ήθελα να αναφέρεται ρητά στο διατακτικό και όρθιο στο αιτιολογικό του κειμένου. Όπως ζητάει το Συμβούλιο. Ξέρετε, όταν ε, ζητάει το Συμβούλιο είτε να, διαγραφούν, να απαλληφθούν είτε να μετακινηθούν στο αιτιολογικό τμήμα οι, κάποιες διατάξεις, πάντα είμαι πολύ επιφυλακτικός, ξυπνάνε υποψίες. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτή την υπόθεση και στη γραμμή που ακολουθεί το Συμβούλιο προ τι δικές μου θέσεις ιδιαίτερα. Μελέτησα κάποιες τροπολογίες των κυρίων, της κυρίας Μπλάστο και του κυρίου Ρικέ. Τη 45 την έχω αποσύρει, αλλά οι 37 και οι 45, ιδιαίτερα οι 37, με δυσκολεύουν. 37 δεν είναι καθόλου σαφή η λογική που επιδιώκει πιο λεπτομερής έλεγχη ξεκινούν μόνο εάν μια αρχική επαλήθευση, ένας αρχικός έλεγχος δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει α, κίνδυνος. Άρα μου λέτε ότι κίνδυνο, ε, πλοίο που παρουσιάζει κανονικό χαμηλό κίνδυνο μπορεί να μην χρειαστεί να ελεγχθεί πολύ λεπτομερώς. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι πρώτα θα έχουμε εντοπίσει ποιο είναι το πλοίο με χαμηλό ή, ή κανονικό κίνδυνο. Δεν καταλαβαίνω ακριβώ που το πάει αυτή η τροπολογία. Στη 44, λέει ο πολιτής. Δεν θα ήθελα να ενισχυθούν οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις σε πλοία. όταν ε, προεξέχοντες παράγοντες ε, και απρόβλεπτοι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν ε, σε μια επιθεώρηση ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα παρελθόν από την τελευταία περιοδική επιθεώρηση του πλοίου, συμπληρωματική επιθεώρηση λόγω μη αναμενωμένων παραγόντων, επαφείται στην επαγγελματική κρίση του υποθεωρητή. Δεν ξέρω ακριβώ ε, τι είδου πρόθεση κρύβεται, ή μάλλον τι είδου αποτέλεσμα μπορούμε να περιμένουμε από αυτή τη διάταξη, αν θέλουμε να περιορίσουμε ε, τι επιθεωρήσει. Αυτέ είναι οι δικέ μου αμφιβολίε. Παρακαλώ του και οδηγητέ τώρα μα δώσουν τι θέσει του. Ο κύριο Κιμουτσάκο, παρακαλώ, από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο ε, και θα ακούσουμε και την κυρία Μάισνερ. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται κανένα άλλο. Και ο κύριο Βαντάλα. Κύριε Κιμουτσάκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η περιγραφή που κάνατε σχετικά με το που βρισκόμαστε σε αυτό το σχέδιο οδηγίας είναι ακριβής. Ε, υπάρχει μεγάλη σύμπτωση απόψεων του ε, κόμματός μας με πολλές από τις τροπολογίες που καταθέσατε, γιατί ο σκοπός είναι κοινό. Μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερη προστασία στους ναυτικούς, μεγαλύτερη ασφάλεια στο πλοίο. Όμως, ταυτόχρονα υπάρχουν και σοβαρά σημεία αποκλήσεων μεταξύ της δικής σας ερμηνείας της κατάστασης και της δικής μας. Δεν είναι απόκληση προς το στόχο. Όπως σας είπα, ο στόχος είναι κοινό, πιστεύουμε τα ίδια πράγματα. Αυτό το οποίο μας κάνει να είμαστε επιφυλακτικοί σε ορισμένες από σας είναι κατά πόσον αυτές είναι πραγματικά εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στην τροπολογία σας νούμερο 2 που είναι το Regression Clause και ενώ επί της αρχής θα μπορούσε κανείς να συμφωνεί βλέπω με δυσκολία πως ένας επιθεωρητής που θα σκούσε τα καθήκοντα του κράτους λιμένος θα μπορούσε πέραν της MLC να έχει βαθιά γνώση και επάρκεια στον τρόπο που μπορεί να γνωρίζει και να εφαρμόζει διατάξεις μιας νομοθεσίας του κάθε κράτους μέλους. Επομένως μπορεί να εισηγούμεθα μια αρχή η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει πολιτική σημειολογία και εκεί αν θέλετε δεν διαφωνούμε αλλά επειδή εδώ μιλάμε για ένα νομικό νομοθετικό κείμενο, δεν βλέπουμε πώς ακριβώς αυτή η αρχή θα μπορούσε να εφαρμοστεί με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Αυτό ως προς την πρώτη παρατήρηση στο βασικό σημείο που αφορά το No Regression Clause. Το άλλο σημείο στο οποίο έχουμε απόκληση είναι ο τρόπος που θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη για να υιοθετήσουν και να κυρώσουν την ε, MLC. Εκεί πάλι συμφωνούμε στον τελικό στόχο. Αναζητάμε όμως ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ενθαρρύνουμε κράτη, το κράτος σημαία να κυρώσει αυτή τη συνθήκη. Και θεωρούμε ότι δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος πλοία τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία ενός εφοπλιστή. Το κράτος του οποίου, το κράτος σημαίας, δεν έχει κυρώσει τη συνθήκη να υφίσταται επιπλέον ε, ε, επιθεωρήσεις όταν ο ίδιος και το πλοίο του είναι άψογο πολλές φορές πάνω από τα στάνταρτς ασφαλείας που χρειάζονται και απλώς θα υφίσταται αυτή την επιπλέον ταλαιπωρία με κόστος σε χρόνο και χρήμα μόνο και μόνο γιατί η κυβέρνηση του κράτους σημαίας δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση. Άλλωστε, στα νιολόγια που αυτά τα πλοία καταγράφονται, όταν το κράτος σημαία δεν έχει κυρώσει τη συνθήκη, αυτό καταγράφεται και στον ιολόγιο. Όταν το πλοίο καταγράφεται στον ιολόγιο. Επομένως εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να επιβαρυνθεί πολύ περισσότερο το, ε, ένας επιχειρηματίας, ένας ιδιοκτήτης, η βιομηχανία, παρά το γεγονός ότι θα τηρεί απαρεκλήτω τι ε, γραμμές ε, της ε, σύμβασης. Τώρα, Όσον αφορά, γιατί βεβαίως δεν πρόκειται να αναφερθώ σε όλα τα, σε όλα τα άρθρα, ε, θέλω να αναφερθώ και στο θέμα ε, του, ε, του χρόνου εφαρμογής. Ε, προτείνεται να αρχίσει να τεθεί σε ισχύ η, η, η οδηγία ένα μήνα μετά την υιοθέτησή της αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο χρόνος, εγώ καταλαβαίνω τον διαπραγματευτικό λόγο για τον οποίο το επικαλείστε, αλλά απ' την άλλη δεν είναι ρεαλιστικός. Είναι αναφυσβήτητα ρεαλιστικότερος ο χρόνος των 18 μηνών, των 12 μηνών ε, που ε, θέτει στην πρότασή της η Επιτροπή. Έχουμε και έναν συνάδελφο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που έχει καταθέσει τροπολογία για 18 μήνες. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι το 12 είναι ρεαλιστικό. Ε, ο ένας μήνας αναφυσβήτητα κινείται πέραν των δυνατοτήτων κάθε κράτους μέλους. Αυτά, ε, αν θέλετε, είναι οι βασικές μας διαφορές. Όσον αφορά στην, ε, ε τροπολογία σας νούμερο 21 που την εντάσσεται στο παράρτημα 10 εκεί πάλι έχουμε σύμπτωση στην φιλοσοφία του πράγματος αλλά θα πρέπει να ξαναδούμε αν αυτά τα οποία καταγράφεται στην τροπολογία σας θα πρέπει να οδηγούν και σε κράτηση του πλοίου είναι ένα βήμα πολύ πιο σοβαρό από τα όσα προβλεπόντουσαν μέχρι τώρα και θα πρέπει να το εξετάσουμε και αύριο θα κοινοποιήσουμε και τη θέση μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να σας. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ήδη όταν είχαμε την πρώτη συζήτηση, ήδη είχα πει ότι εγώ για την ομάδα μου πολλά μπορώ να υποστηρίξω και τα θεωρώ σωστά από αυτά που τροποποιήθηκαν τώρα. Non-regression clause. Δεν τη βρίσκω τόσο δύσκολη και δυσχερή. Είπε ο κύριος Κουμουτσάκος, κανένας δεν μπορεί να ξέρει όλες τις εθνικές νομοθεσίες. Δεν χρειάζεται να το κάνει κανείς αυτό. Πρέπει να ξέρει τι γίνεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία να δούμε αν είναι δυνατόν να υπάρχουν καλύτερες διατάξεις όσον αφορά τους απασχολούμενους, τους εργαζόμενους σε σχέση με την ανώτερη θέση στην οποία βρίσκεται ανέβει το ευρωπαϊκό δίκαιο έναντι του εθνικού δικαίου. Και αυτό δεν είναι τίποτα το δύσκολο ή τρομερό, διότι αν υπάρχει ένα εθνικό δίκαιο το οποίο είναι αυστηρότερο, τότε αυτό δεν απαγορεύεται και στην οδηγία, την ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο και κάτι τέτοιο ε, μπορεί να προβλέπεται και που πολλές φορές δημιουργεί για τη Γερμανία ένα ειδικό πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα για την ομάδα μας εμείς. Για τα πλοία, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κουμουτσάκος το κατανοώ, οι πλειοκτήτες ε, υφίστανται κυρώσει, ε, οι οποίοι φέρθηκαν σωστά και συμμορφώθηκαν ενώ το κράτος του είναι εκείνο το οποίο δεν κινητοποιήθηκε σε σχέση με την επικύρωση και όταν θα έχει γίνει, όταν θα γίνει αυτό, θα είναι ένα κίνητρο, διότι οι πλειοκτήτες θα καταβάλουν προσπάθειες ήδη στη χώρα τους ε, για να υπάρξει αυτή η προσαρμογή, αυτή η συμμόρφωση με αυτή την επικύρωση. Και ούτε και εδώ θα βλέπα να υπήρχαν προβλήματα. Δηλαδή ουσιαστικά σε πολλά πράγματα μπορώ να συμφωνήσω με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Βαντάλεν. Βαντάλεν παρακαλώ. Δεν θέλει ο κύριος Βαντάλεν. Καλώς. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις επικοδομητικές αυτές τροπολογίες. Από πλευράς της Επιτροπής προς είναι αποδεκτές. Δώδεκα μας δυσκολεύουν κάπως μεταξύ των οποίων οι τροπολογίες του ΕΛΚ που αποδυναμώνουν αυτό που στην αρχική μας ε, πρόταση θεωρούσαμε ότι θα ενισχύει το ρόλο του κράτους του Λιμένα για τις επιθεωρήσεις με ένα πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού για τον κλάδο. Ρήτρα δηλαδή, τη ρήτρα δηλαδή, βάσει της οποίας το πλοίο σημαία χώρας που δεν έχει κυρώσει την σύμβαση θα υπάρχει πάγεται σε περισσότερες επιθεωρήσεις. Δηλαδή, ζητούν τα κράτη-μέλη να κυρώνονται βέβαια οι συμβάσεις και αυτή η διάταξη, αυτό που θα κάνει είναι ότι θα δώσει κίνητρα προς τα κράτη, αρχική δηλαδή διάταξη, ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους από, προς την IMO. Για δε την αρχική πρόταση που είχαμε εμείς εισαγάγει με το άρθρο, ύστερα από μια νέα διατύπωση, για να ακολουθήσουμε τις θέσεις σας, στο να παραμένει το σημείο αυτό ως άρθρο και να μην πάει στο αιτιολογικό, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο αρμόδιος από πλευράς του λιμένος θα δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα το κράτος της σημαία πρέπει να μεριμνεί ώστε τα πάντα να είναι εντάξει. Για τις λοιπές τροπολογίες. Οι τροπολογίες ιδιαίτερα υπαριθμών 3, 4, 36 και 37 μας γεννούν κάποιες δυσκολίες γιατί ανατρέπουν τη λογική του ελέγχου από το κράτος του λιμένου, που σημαίνει ότι ο επιθεωρητής ανεβαίνει στο πλοίο, κάνει τον έλεγχο στα χαρτιά, κάνει μια πρώτη επιθεώρηση επισκεπτόμενο στο πλοίο. Εάν δεν βλέπει κανένα πρόβλημα, τελειώνει η ιστορία. Εάν δει ότι χρειαστεί, προχωρεί σε πιο λεπτομερή επιθεώρηση και καταγράφει ελλείψεις. Με τις τροπολογίες λοιπόν που σας ανέφερα, στο πλαίσιο της MLC ε, βλέπουμε ότι να πηγαίνουν υπερβολικά μακριά, ιδιαίτερα η 33 που τίνει να επεκτείνει τον ε, έλεγχο του κράτους λιμένος, λιμένος υπογραμμίζω, σε όλα τα πλοία και πληρώματά του σε ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του κράτους Μαλουλές, Στα εγχώρια ύδατα. Αυτό είναι υπερβολικό και μάλιστα μη εφικτό. Επίσης, Όπως επεσήμανε και ο κύριος Πρόεδρος, ο συζητητής, υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες ε, είναι κάπως ακραίες, όπως η 44 που αναφέρεται στο θέμα της μη κύρωσης ως λόγου, ειδικού λόγου για επιθεώρηση. Αυτό σημαίνει ότι το, το πλοίο μετατρέπεται σε κινούμενο στόχο για κάθε επιθεωρητή ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό, δηλαδή να ε, μπουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους τα σκάφη των οποίων ε, το κράτος σημαία δεν έχει επικαιρώσει κάποια διεθνή σύμβαση. Μια άλλη τροπολογία που θέλω να επισημάνω ήταν η παριθμόν 41 που σχετίζεται με την πρόσβασιμότητα, τη δυνατότητα πρόσβαση όλη πληροφορία δεδομένων των επιθεωρήσεων. Πρόσβαση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. από τι αρχέ ελέγχου του κράτου λιμένα πρέπει να προσφέρετε πρόσβαση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε να σα πω, αυτά όλα υπάρχουν στην ιστοσελίδα τη Ευρωπαϊκή ε, υπηρεσίες για την ασφάλεια των θαλασσιών μεταφορών σε πρώτη βάση. Ένα δεύτερο επίπεδο πληροφόρησης ε, υπάρχει, πληροφορίες μάλλον υπάρχει, στη διάθεση του επαγγελματία ή του επιθεωρητή στους λιμένες. Όχι. Στη δική, δεν είναι ανοιχτό στη δική μας πρόσβαση οποιοδήποτε άλλο. Έχει να κάνει με λεπτομερεί πληροφορίε, προ το πότε έφτασε το σκάφο, τι ε, φορτίο μεταφέρει, εάν πρέπει να πρόκειται να υποβληθεί σε επιθεώρηση, αν έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση, όλα αυτά ε, διαθέσιμα σε πιο περιορισμένο κύκλο προσώπων από τις αρχές. Αλλά όπως είπα, το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει πληροφορίες στη διάθεσή του αντίστοιχες με αυτές που ε, διαθέτει και το Συμβούλιο εξού και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την τροπολογία. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Για να απαντήσω μόνο, να σας πω για αυτή τη ρήτρα non-regression αν και η κυρία Μάισνερ ε, απάντησε όσο καλά θα μπορούσα να σας απαντήσω κι εγώ. Αν δεν υπάρχει αυτή η ρήτρα, τότε θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικές προδιαγραφές και εμείς ουσιαστικά λέμε ότι εντός των ευρωπαϊκών σκαποφών ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάρχει εργασιακό δίκαιο το οποίο εφαρμόζεται και αυτό ακριβώς ε, προϋποθέτει αυτή η ρήτρα non-regression. Τώρα, για τα κράτη σημαία που δεν κυρώνουν. Εάν ένα κράτος σημαίας δεν κυρώσει τη συνθήκη, τότε το κράτος σημαίας δεν θα κάνει ελέγχους βάσει της σύμβασης. Αφόσον δεν το κυρώνουν, τότε ε, δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έλεγχο. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μεγαλύτερο κίνδυνο μη συμμόρφωσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν κάποιοι από εμά λοιπόν θεωρούν ότι και τα 27 κράτη-μέλη έχουν το πιο εξαιρετικό σύστημα για τις θαλάσσιες μεταφορές ε, και για τις συμβάσεις ε, ναυτικής εργασίας, ε, τότε μάλλον να πατάστε εκτρά έχουμε κράτη-μέλη τα οποία είναι μαυροπινακισμένα και βρίσκονται και στα χειρότερα μνημόνια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα πάντα είναι ρόδινα λοιπόν στον Ευρωπαϊκό Παράδεισο.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 Ακούγεται τώρα. Ακούγεται τώρα κύριε Κουμουτσάκο. Also dieser Vorschlag Αυτή η πρόταση ευθυγραμμίζεται με την προηγούμενη. Αφορά τη συμφωνία του 2006 όπου οι διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων για πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενους ε, ναυτικούς και Ξέρουμε ότι η αρμόδια είναι η Επιτροπή Απασχόλησης ΕΜΠΛ. Με αυτή την οδηγία οι ευρωπαϊκές διατάξεις ε, με τους τίτλους 1, 2, 3, 4 ευθυγραμμίζονται που καθορίζονται τα δικαιώματα των ναυτικών. Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι που τη συμφωνία τους αυτή μέσω μιας απόφασης του Συμβουλίου θέλουν να την υλοποιήσουν σε σχέση με αυτή την συμφωνία στον τίτλο 5 για την ένταξη αυτών των θεμάτων επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τα αναγκαία βήματα και διαβήματα για να ε, τα εντάξει σε ένα κοινό πλαίσιο. Από τις 37 τροπολογίες ε, κατατέθηκαν περαιτέρω 7 που μπορώ να συμφωνήσω χωρίς ε, επιφυλάξεις. Έχω ένα πρόσημο συν θετικό για την, ε, τον πίνακα ψηφοφορίας. Επιπλέον τη δική μου τροπολογία 3 την αποσύρω. Το αποφάσισα αυτό για λόγους ε, συνεκτικότητας και συνοχής και την τροπολογία 4 επίσης και αυτή αποσύρεται διότι η τροπολογία 41 από πλευρά συναδέλφου Φλέκενστάιν είναι πιο ολοκληρωμένη από πλευρά διατύπωση. Επαρκούμε σε αυτά τα σχόλια. Θα περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σα. Προσδοκώ να τα ακούσω. Ευχαριστώ. Από του σκιώδη είσαστε ο μόνο παρόν. Θέλετε να πείτε κάτι εσεί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρόκειται για τη συμφωνία για τους ναυτικούς να υπάρξει μια αντιστοίχηση εδώ η αρμόδια τη ουσία είναι η Επιτροπή Απασχόληση, ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Έχω κάποιε μικρέ αμφιβολίε αν όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν εδώ έτσι όσο έχουν. Πολλά μπορώ να τα τονίσω και να τα υπογραμμίσω για τα Emerging Labor Certificates, τα πιστοποιητικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπογράφουν τα κράτη-μέλη. Αν αυτό το συμπεριλάβουμε στο ευρωπαϊκό δίκαιο δεν θα είναι διπλοεπικάλυψη. Είναι αναγκαίο να γίνει αυτό. Είναι θέμα επικουρικότητας είναι σαφές. Εκείνος ο οποίος υπογράφει πρέπει να ε, ευθυγραμμίζεται και να συμμορφώνεται σε σχέση με τις συμφωνίες για τους ε, εργαζόμενους στη θάλασσα, για τους ε, ναυτικούς και για τις, τη διαδικασία των procedures ήδη προβλέπεται και υλοποιείται στο ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει εδώ να επαναληφθεί αυτό αφού υπάρχει ήδη και, και λειτουργεί. Είναι μια ε, διπροεπικάλυψη. Κατά τα άλλα συμφωνώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλατε εσείς να πείτε κάτι πολύ σύντομα, 20 δευτερόλεπτα να σχολιάσετε. 10 δευτερόλεπτα χρειάζομαι μόνο γιατί ο Κνούτ, ο σκιώδης εισηγητής μας ζήτησε να πω ότι ακολουθεί τις απόψει του εισηγητή απόλυτα. Υποστηρίζει τη θέση του εισηγητή. Δεν θα υπάρχουν προβλήματα λοιπόν από την ομάδα μα σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσείς. Μια πολύ σύντομη αποσαφήνιση, διευκρίνηση σε σχέση με, για την τροπολογία 12 τώρα πραγματικά τίθεται το ερώτημα. Αυτό δεν διπλοεπικαλύπτει το άρθρο 3 στην πρακτική εφαρμογή και δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί σύγχυση για το ποιε προδιαγραφέ θα πρέπει να υλοποιούνται. Παρακαλώ ο εισηγητή να προβληματιστεί, να δει τι συμβαίνει εδώ και πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τροπολογία 12. Μπέρκ παρακαλώ. Μπορείτε να είσαστε σύντομοι κι εσείς. Ε, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και θα πω στον αρχηγό σας ότι ε, από πλευρά σας υπήρξε ο πρόσθετος χρόνος. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Νομίζω το μεγαλύτερο ζήτημα αφορά την έκδοση ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού επιπλέον πέρα από το διεθνές πιστοποιητικό MSC όπου βλέπουμε να υπάρχει διπλή υποχρέωση από τα κράτη-μέλη, διπλή επιβάρυνση. Γι' αυτό για τις τροπολογίες 2 και 6 δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από εμάς. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι με την τροπολογία 38 ένα νέο εδάφιο, ένα νέο σκεπτικό εισάγεται σε σχέση με αυτή την οδηγία που προτείνεται να αλλάξει. Το MLC θα εξαιρείται από τις άλλες συμφωνίες όπου το κράτος σημαίας ε, θα έχει ε, δικές του διατάξεις ε, σε σχέση με την αξιολόγηση ποιότητας. Το MLC δεν θα πρέπει λοιπόν ξεχωριστά σε σχέση με τις άλλες συμφωνίες να μπορεί να λειτουργεί. Αυτό δεν θα το δεχόμασταν. Για τα άλλα, για το θέμα το οποίο προηγούμενα αναφέρθηκε, για την τροπολογία 12, που θα μπορούσε να δημιουργεί διπλοεπικάλυψη, δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη ξεχωριστή δυσκολία με αυτό. Δεν νομίζουμε να υπάρχει αντίφαση σε αυτό. Αυτό σε σχέση με τα σχολεία μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιώργο εσύ. Euh, Ευχαριστώ. Θα έλεγα τα δύο αυτά σημεία που από πλευρά τη συναδέλφου Μάισνερ αναφέρθηκαν νομίζω θεμητό είναι αλλά αυτό που θέλαμε εμείς είναι πρώτον τα κράτη-μέλη να μην απαιτείται να εργάζονται με διαφορετικά έγγραφα, να είναι ένα συνεκτικό και ας το πω έτσι ε, αποτελεσματικό έγγραφο που να μην δημιουργεί κάποια επικάλυψη. Είναι απλούστερο στη συνέχεια με ένα πλήρες έγγραφο να μπορεί να εργάζεται κανείς, ολοκληρωμένο έγγραφο, αντί ε, εμβαλωματικά να μπορεί να πρέπει να το χρησιμοποιεί ή να το υποβάλει. Εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να πω ότι τις ε, επιφυλάξεις αυτές ε, και για τα πιστοποιητικά θα ήθελα να παραμείνω στις δικές μας ε, απόψεις και θέσεις. Ευχαριστώ. πρόεδρο. ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε αύριο και αυτό το θέμα. Καταφέραμε να επανέλθουμε έγκαιρα, Γιώργο, εσύ και εγώ μεταξύ μας και τώρα προχωράμε στη συνάντηση των συντονιστών σε δύο λεπτά. Όσοι δεν θα συμμετάσχουν να αποχωρήσουν παρακαλώ.